Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Έχουμε ακόμη ένα φορτωμένο πρόγραμμα για σήμερα το απόγευμα. Να μην καθυστερήσουμε λοιπόν ιδιαίτερα. Στο σημείο 30. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτησή μας ε, σχετικά με την έκθεση του Ρίτσαρτ Χάουιτ για μια δημόσια κρέωση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και πορεία πιο μιας βιώσιμη ανάκαμψη χωρίς αποκλισμούς Όπως ε, γνωρίζετε, στο πλαίσιο αυτό Έχουμε μια ανταλλαγή με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων που επίσης ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό και τελικά θα έχουμε μια διασταύρωση μεταξύ δύο εκθέσεων πρωτοβουλίας και έτσι θα συνεργαστούμε. Όμως σήμερα ο στόχος μας δεν είναι να εξετάσουμε το κείμενο του κυρίου Χάουιτ, αλλά να ακούσουμε τους προσκεκλημένους μας που παρευρίσκονται εδώ στα δεξιά σας και στα αριστερά μου. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Χάουιτ να κάνει μια εισαγωγή για τη συζήτηση και κατόπιν να δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους μας για να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους και θα έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις. Παρακαλώ κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, για τα εισαγωγικά σας σχόλια και για την προσωπική σας υποστήριξη για το θέμα αυτό. Ξέρω ότι η εταιρική ευθύνη είναι κάτι που σας έχει απασχολήσει και εγώ εκτίμησα τις συμβουλές σας. Νομίζω ότι για τέταρτη φορά είχα την τιμή να είμαι εισηγητής για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ελπίζω ότι έχω συνεισφέρει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συνεισφέρω σε αυτό το έργο. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία για την υποστήριξή της. Σήμερα το απόγευμα έχουμε μια δημόσια κρόαση γιατί ήθελα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής και όσους παρακολουθούν το έργο μας να κατανοήσουν σε σχέση με την τελευταία ανακοίνωση Κομισιόν που είχαμε πριν πέντε έτη ότι πολλά έχουν αλλάξει. Πολλά έχουν αλλάξει στη νέα ανακοίνωση και ήθελα να καλωσορίσω τη νέα ανακοίνωση δημοσίως γιατί ε, νομίζω ότι αποτελεί ένα θετικό και βήμα και μια επικοδομητική βάση για να προωθήσουμε την πολιτική στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στα ευρωπαϊκά όργανα. Και κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι η συζήτηση μεταξύ των επιχειρήσεων και από τις επιχειρήσεις και με τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει πολύ διαφορετικό ύφο σήμερα σε σχέση με πέντε έτη πριν. Ορισμένα μέλη της Επιτροπής ε, ήταν ε, και στο Κοινοβούλιο και στην τελευταία έκθεσή μου είχαμε ε, κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμβασμό τελικά, αλλά δεν ήταν εύκολο και δεν ήταν εύκολο στο κύριο όργανο που προωθεί την πολιτική αυτή στις Βρυξέλλες, ε, το Φόρουμ των Stakeholders των Διαφερομένων Μερών. Προσωπικά είχα εκεί ε, την τιμή να προσωπώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως είχαμε μία περίοδο που αποχώρησαν οι ΜΚΟ από το Φόρουμ και δεν εργάζονταν ε, ενεργητικά. Όμως ε, τώρα είναι διαφορετική η κατάσταση και ξέρω, το ξέρω αυτό και θέλω να το καταλάβουν αυτό όλοι οι φίλοι ε, στην Επιτροπή. Το Φόρουμ συνεργάζεται εδώ αποτελεσματικά στις Βρυξέλλες τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Έχει μετακινηθεί και η Κομισιόν και είπε ότι θέλει μια ανοιχτή στρατηγική και αυτό διευκολύνει την ε, νέα συνένεση και έχει δοθεί μια νέα όθηση, μια νέα ενθάρρυνση σε αυτό το τομέα πολιτικής. Όμως κάτι άλλο που έχει αλλάξει είναι στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών όπου αυτά τα θέματα για την εταιρική ευθύνη ε, συζητώνται σε παγκόσμιο επίπεδο και πάλι εκεί υπήρχε μεγάλη πόλωση. Επικεντρώθηκαν στι συζητήσεις ε, που αφορούσαν τις επιχειρήσεις και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα εργατικά δικαιώματα και ε, Επίση, πριν 5-6 χρόνια ε, και δεν ήταν σε μια ιδιαίτερα απολωμένη θέση, όμως ε, ο ειδικό ε, εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών είχε αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο και κατόρθωσε να οδηγήσει σε συνένεση και μπορώ να πω ότι υπήρξε ένα πολύ αρνητικό κλίμα, μια πολύ αρνητική συζήτηση και έδειξε ότι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχουν υποχρεώσεις που βασίζονται στην νομοθεσία του Σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι κυβερνήσεις και οι εταιρείε έχουν νομικές υποχρεώσεις. Ε, βέβαια αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε να το συζητάμε σε καμία περίπτωση. Αλλά επίση μπόρεσε να βρει και έναν τρόπο να προχωρήσουμε και έκανε ένα έξυπνο μείγμα ρύθμιση ε, και εθελοντισμού. Και έτσι υπήρξε η υποστήριξη των επιχειρήσεων στο σύστημα του ΙΕ. Και η Ένωση των ε, εργοδοτών και τα ε, διεθνή εμπορικά επιμελητήρια όπως ε, και οι ΜΚΟ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπόρεσαν να υποστηρίξουν το έργο αυτό. Και θέλω να πάρω αυτή τη νέα όθηση, να αντιβάλλω στον τρόπο με τον οποίο συζητάμε αυτή την έκθεση εδώ στο Κοινοβουλίο και με το συνάδελφο τον κύριο Μπαλτασάρη στην Επιτροπή Νομικών Θυμάτων. Σκοπεύουμε να συνεργαστούμε πολύ στενά, είχαμε πολλές παράλληλες συζητήσεις και απευθύνομαι στους σκιώδεις και σε όλους ε, που συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή να σκεφτούμε ένα ε, νέο συμβιβασμό, τη νέα συνένεση που υπάρχει γύρω από την εταιρική κοινωνική ευθύνη και προκειμένου να το προωθήσω αυτό. Τι κάναμε με την ακρόαση σήμερα το απόγευμα. Καλέσαμε τρει ομιλητέ που εκπροσωπούν τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, τα συνδικάτα, τι επιχειρήσει και τι ΜΚΟ Έχουμε και την Nova Nordisk, ε, συμμετείχε στο Ρίο στην Σύνοδο για την αηφόρο ανάπτυξη. Εκεί πολλές εταιρείε ήθελαν να συζητήσουν τις δικές τους δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη. Και η Novo Nordisk είναι μία από τις ε, ε που ήταν ε, εκεί τις κύριες επιχειρήσεις ε, και με την Ένωση Επιχειρήσεων που συμμετείχε από την Ευρώπη. Υπήρξε μεγάλη συνεισφορά σε αυτή τη συζήτηση. Ίσως ε, λοιπόν ε, κάποιοι που δεν γνωρίζουν τόσο καλά το ζήτημα το να ακούσουν την συνεισφορά της Nova Nordisk σε αυτόν τον τομέα θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια άποψη για το τι μπορεί να γίνει. Εγώ πιστεύω ότι αποτελούν ένα πολύ καλό παράδειγμα και καλωσορίζω το γεγονός ότι έχουμε εκπρόσωπό τους εδώ. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, Έχουμε εδώ τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον ξέρω για πολλά χρόνια και έχει ασχοληθεί με την υφαντουργία και ασχολείται με τις καταχρήσεις ε, στη ε, αλυσίδα του εφοδιασμού, με τις κακές συνθήκες εργασίας, ε, με την παιδική εργασία και νομίζω ότι αυτή η Ένωση ήταν η κύρια Ένωση που ασχολείται με αυτά τα θέματα της εταιρική κοινωνικής ευθύνης και στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Και τώρα έχει αναλάβει την ε, θέση τον πληρωθεί Γενικού Γραμματέα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Συνδικάτων. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Μερικές φορές είναι δύσκολο για τα συνδικάτα να μπουν σε αυτή τη συζήτηση με όλες τις προτεραιότητε που έχουν. Όμως νομίζω ότι θα είναι πολύ θετική η συνεισφορά του. Και τέλο έχουμε τον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό για την εταιρική δικαιοσύνη είναι μια ομάδα ομπρέλα και εκπροσωπούνται 30 οργανώσεις από την κοινωνία των πολιτών και ε, εκεί οδηγούνται από το δίκτυο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Ευρώπη που διερευνά ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση έτσι λοιπόν έχουμε κάποιου πολύ σημαντικού εμπειρογνώμονε που θα μπορούσαν να μα ενημερώσουν για το τι συμβαίνει σε αυτό το τομέα πολιτική και θα σκεφτούν μαζί μα ε, για την ανακοίνωση τη Κομισιόν. Με αυτή την εισαγωγή θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου γιατί θέλω να του ακούσω. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν αμφισβητούμε καθόλου ότι θα μας διαφωτίσουν επί των προτάσεων της Κομισιόν. Έτσι λοιπόν, θα τους δώσω δυστυχώς ε, το λόγο για πέντε λεπτά Ξέρω ότι είναι λίγος ο χρόνος, αλλά αυτό διαθέτουμε. Και θα ξεκινήσουμε από την κυρία Ελίνα Βρόντσκι, που είναι πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού για την Εταιρική Δικαιοσύνη. Και φαντάζομαι ότι θα την έχετε συναντήσει ήδη στα πλαίσια εξέτασης διαφόρων άλλων φακέλων. Πρόκειται για μια οργάνωση που κάνει εξαισιομία τη δουλειά και για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα. Έχετε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα εξ ονόματος ε, της ε, Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ε, για την εταιρική δικαιοσύνη να σας μιλήσω καταρχήν για το νέο ορισμό που έχουμε δώσει. Αυτός ο νέος ορισμός υπάρχει στην ανακοίνωσή μας, στα πλαίσια βέβαια της νέας οδηγίας, όπως είπε ο κύριος Χάουιτ, αλλά και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ. Η δήλωση αναγνωρίζει ότι βεβαίως οι εταιρείες έχουν και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, είναι υπεύθυνε και βεβαίως από εκεί και πέρα μπορεί να ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση για την εθελοντική και υποχρεωτική τους δράση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι αρνητικές συνέπειες της επιχειρησιακής δράσης μπορεί να δημιουργήσουν ανησυχίες, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και ε, παντού στον κόσμο. Θα σας δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Μία εταιρεία στο Πακιστάν πήρε φωτιά πρόσφατα χάθηκαν πολλές ζωές εργαζομένων και βεβαίως από ό,τι φάνηκε τα μέτρα που είχαν ληφθεί δεν ήταν αρκετά. Το θέμα της ε, Ευρωπαϊκής Εταιρείας, το θέμα της προστασίας των μέτρων ασφάλειας είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη καθώς και το πώς θα μπορούσαν να συνεισφέρουν οι ίδιοι εργαζόμενοι σε αυτός έτσι να αποφευχθούν παρόμοιες ε, περιπτώσεις στο μέλλον και τραγωδίες. Βλέπουμε βεβαίως ότι παρόλο που σήμερα υπάρχουν πολύ θετικές επιπτώσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι προφανείς για τις ίδιες τις εταιρείες, οι κανόνες για την ε, εταιρική διακυβέρνηση και η εταιρική ευθύνη είναι κάτι που σαφώς φαίνεται σε πολλές από τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παραδείγματος χάρη αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από μερικούς μήνες για την κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση. Βλέπουμε ότι υπάρχει δέσμευση από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμοστούν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές και αρχές και αν αυτό βεβαίως δεν είναι αυτός σκοπός, η έλλειψη ενό μηχανισμού επιβολής τους είναι κάτι που σαφώς δείχνει αδυναμία σε διεθνές επίπεδο, χρειάζονται τρόποι να μετρηθούν η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα βελτίωσης αυτών των ρυθμίσεων και την ίδια ώρα να εντοπιστεί τρόπος να παιχθεί ένας ηγετικός ρόλος όπως ε, αυτό που κάνει τώρα η Επιτροπή. Οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές καθώς και η εφαρμογή τους είναι κάτι στο οποίο ξεκίνησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις διαβουλεύσεις και σαφώς θα έχει ε, επιπτώσεις και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρειάζεται μια ανάλυση της συνοχής, της πολιτικής, των αδυναμιών, των κενών, το ίδιο όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις, την εμπιστοσύνη, τη στήριξη στις επιχειρήσεις, κάτι που θα πρέπει να γίνει και να ειδωθεί στα πνεύμα και στο πλαίσιο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. Χρειάζεται ένα, σχέσιο, ένα σχέδιο δράσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει ιδιαίτερα να εξετάσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη για αυτούς που πλήττονται. Επίσης, διαδικασίες ταχείες με τις οποίες μπορούν οι επιχειρήσεις να προσφύγουν όπως αυτό που προβλέπει στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών ο κανόνας για τη σωστή διακυβέρνηση και φυσικά εμείς χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κατευθυντήριες γραμμές για τρεις συγκεκριμένους τομείς. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι μέτρα θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ληφθούν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις άλλες διαδικασίες. Εμείς θεωρούμε ότι η μελέτη που θα δημοσιευθεί που στο, πριν το τέλος αυτού του χρόνου θα περιλαμβάνει και άλλες κατευθυντήριες γραμμές για τον τομέα αυτό. Στηρίζουμε βεβαίως το σχέδιο νομοθεσίας και ελπίζουμε ότι αυτό το σχέδιο θα βοηθήσει τις εταιρείες να αξιολογήσουν συνέπειες και κινδύνους έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιολογήσουν πιο σωστά τους κινδύνους αυτούς. Τελειώνοντας, θα ήθελα να μιλήσω για την πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη. Λυπόμεθα γιατί το θέμα αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στην δήλωση αυτή και ζητούμε από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ακόμα σήμερα τα θύματα καταχρήσεων Θεωρούμε ότι η μελέτη στο Εδιμβούργο που ζητήθηκε πριν από λίγα χρόνια και έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει πολύ σωστές προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο δεύτερος εμπειρογνώμων Πατρίκ Ιτσέρτ, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ειδικό για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ και εξ ονόμου τη Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και τον Ρίτσαρτ. Ο τίτλο ε, τη επόμενη έκθεση είναι φιλόδοξο. Ε, Όμω, ε, είναι πεπισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν θέλει να βγει από την κρίση πρέπει να ληφθεί μια σειρά μέτρων. Τα έχουμε συνοψίσει στο κοινωνικό σύμφωνο και ε, φυσικά η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει θέση εκεί. Για να φτάσω στην ανακοίνωση θα έλεγα ότι το 2006 για μας ήταν εντελώ άδειο το ποτήρι. Σήμερα πράγματι χαιρόμαστε με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και στο μισογεμάτο ποτήρι θα έβαζα και τον νέο ορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πιστεύω ότι κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος, αναφερόμαστε στην, ε, ε, στον ορισμό αυτό και στην ευθύνη των εταιριών σε σχέση με τα άμεσα ή έμεσα αποτελέσματα που επιφέρουν στην κοινωνία και μιλάμε για τη λογοδοσία επιλέγοντας αυτόν τον ορισμό ξεπερνούμε αυτή την ε, συζήτηση που μας ε, δηλητηρίωσε στο φόρουμ των ενδιαφερομένων μερών ε, της ρύθμισης έναντι του θελοντισμού χρειάζεται ένα μείγμα και των δύο για μας είναι σημαντικό ο νέος ορισμός επαναπλησιώνει τη συζήτηση γιατί έχουμε κατανομή των ρόλων πρέπει να προστατεύσουμε την κυβέρνηση να συμβαστούμε τις επιχειρήσεις και κατά να διορθώσουμε και σε άλλες πτυχές τη ανακοίνωση υπάρχει και αναφορά στα διεθνή μέσα, αν και χρειάζεται κάποια ιεραρχία. Όμως ε, γίνεται αναφορά καταρχήν ε, στις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΕ και του ΟΣΑ και για μας ήταν ουσιαστικό. Να υπογραμμίσω επίσης ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη και ε, αφορά ε, και ο σεβασμός ε, των συμβάσεων αποτελεί προαπαιτούμενο και πολλές φορές υπήρξε ένα pick and choose που μας ε, εξέπλητε. Μία φράση που ήταν σημαντική για μας είναι ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνικός διάλογος αλληλοσυμπληρώνονται, αλληλοεμπλουτίζονται. Είναι κάτι που το 2004 δεν μπορούσε κανείς να το γράψει καν. Κανείς δεν να τα ακούσει. Έχουμε σημειώσει πρόοδο το γεγονό ότι η νέα ανακοίνωση αναφέρεται στον άμεσο και μέσο αντίκτυπο στην λυσίδη είναι σημαντικό και επίσης ένα πρόγραμμα εργασίας. Νομίζω ότι το χαιρετήσαμε και αυτό. Λαχθέντος αυτού, το ποτήρι παραμένει για μας μίσο άδειο, γιατί την έχουμε ένα πρόγραμμα εργασία, καλό είναι, αλλά φυσικά πρέπει και να τεθεί σε εφαρμογή. Έτσι λοιπόν στην υλοποίηση Πολλά θα έπρεπε να γίνουν πριν τα τέλη του 2012 και θα αναφερθώ συγκεκριμένα στη δέσμευση της Κομίσιον να δημοσίευσει πριν τα τέλη του 2012 μία έκθεση για τις προτεραιότητες της Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κατητηρίων αρχών των Ηνωμένων Εθνών και κατόπιν ε, να δημοσιεύει προοδευτικές εκθέσεις. Πρέπει η Κομισιόν να δώσει το καλό παράδειγμα. Δεύτερον, η Κομισιόν επίση δεσμεύτηκε να παροτρύνει τα κράτη-μέλη να, ε, να καταρτήσουν εθνικά σχέδια εφαρμογή πριν τα τέλη του 2012. Και είχαμε ένα καλό παράδειγμα στη Δανία, αλλά υπάρχει μία σειρά άλλων χωρών ε, όπου υπάρχουν ερωτηματικά. Τρίτον, έχουμε τι επιχειρήσει. Ε, το συζητήσαμε και αυτό προηγουμένω. Αλλά όταν η Κομισιόν λέει ότι περιμένει τις επιχειρήσεις ε, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ίσως ε, μιλάμε εδώ ότι περιμένουμε τον κοντό. Μπορεί και να απογοητευτούμε. Τέταρτον. Η Κομισιόν ε, δεσμεύτηκε πριν τα τέλη του έτους να, υπογράψει, να παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση για τη διαφάνεια των πληροφοριών ε, σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε από τη διαφάνεια και η έκθεση αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί μέσω των επιτροπών, των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει αλληλοεμπλουτισμό. Ε, και σήμερα υπάρχουν κάποια δισταγμοί και ότι μπορεί να καταλήξουμε σε κάτι soft, δηλαδή κάτι μισκόπιμο. Θα ήταν λάθος να περιμένουμε Ήδη πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει πλαίσια, δεν θα περιμένουμε και 27 να αποκτήσουν ένα πλαίσιο για να προβούμε στην ε, ενοποίηση. Τώρα πρέπει να το κάνουμε. Οι μικρές και μισές επιχειρήσεις ε, διαφέρουν. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε ορισμένες ιδιαιτερότητε των ΜΜΕ, αλλά όχι επί της αρχής, δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε παιδική εργασία με μικρές και μεσές επιχειρήσεις, αλλά σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να υπάρχει απλούστευση, αλλά είμαστε αντίθετοι σε αυτή την ιδέα να αποκλειστούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η προηγούμενη ακρόση ανέφερα κάτι το αληθές πριν κάποια χρόνια όταν κατέρευσε ένα εργοστάσιο στον Μπαγκλαντές. Λυπούμε που το λέω, αλλά μία από τις επιχειρήσεις ήταν βελγική. Και ήταν ε, ένα γραφείο με δύο άτομα στις Βρυξέλλες και τίποτα άλλο δεν έκανε παρά αντίστροφες δημοπρασίες. Ήταν ο κύριος ε, δηλαδή με τη γραμματεία του γραφείου, του έφταναν ε, κάποιες παραγγελίες και από την άλλη έκανε κάποια τηλεφωνήματα στο Παγκλαντές και ουσιαστικά έκανε κοινωνικό ντάμπινγκ χωρίς να τον ενδιαφέρει. Και αν ε, είχαμε ε, κάνει υποβολή εκθέσεων θα καταλαβαίνουμε ότι είχαμε μεγάλο τζίρο και ουσιαστικά με υπεργολαβή απασχολούσε πάρα πολλά άτομα. Τώρα, ε, για τις δημόσιες προμήθειες δεν νομίζω ότι επειδή είναι η κρίση πρέπει να εγκαταλείψουμε το στοιχείο αυτό και θα πρέπει και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια να είναι στο ίδιο επίπεδο. Επίση, αναφερθήκαμε στι ε, ε, απατηλέ εμπορικέ πρακτικέ. Μιλάμε για το greenwashing. Μα ανησυχεί κάπω η ιδέα τη Κομισιόν να βάλει μια τιμή. Καλό είναι αυτό, αλλά πριν ε, κάποια χρόνια βρήκαμε ένα pick and choose, δηλαδή μια δυνατότητα επιλογής και ε, μπορώ να σας πω ότι υπήρξε θέμα με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η τερκή κοινωνική σχέση πρέπει να εισαχθεί σε όλες τις πολιτικές, στην εμπορική πολιτική, το είπε και ο Ρίτσαρτ. Ε, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στις ευρωπαϊκές συμφωνίες πλαίσιο και στις διεθνείς συμφωνίες πλαίσιο και στο δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης θα υπάρξει και ένα ψήφισμα που θα περάσει από την επόμενη εκκληστική επιτροπή μας την επόμενη εβδομάδα και εκεί υπάρχει σαφής τοποθέτηση υπέρ ενός πλαισίου ε, επιλεκτικού για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Εγώ που πιστεύω προσωπικά ότι έχουν προκύψει πολλά από αυτό Τώρα, ε, πρέπει να έχουμε λοιπόν την προσέγγιση με τα διαφορεμένα μέρη. Δεύτερον, διαφάνεια, υποβολή εκθέσεων. Ε, σήμερα ε, μιλάμε για μια αγορά 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή για πολύ μεγάλες ε, ε συναλλαγές. Στο Κόλμη το 2009 η καλύτερη έλεγχη ήταν να υπάρχουν ελεύθερα και να ανεξάρτητα συνδικάτα. Τρίτον, το είπαμε ότι ε, την ε, ιατρική κοινωνική ευθύνη. Έχουμε, έχει περάσει σήμερα στις 20.000. Ε, νομίζω ότι δεν έχουμε σήμερα πολύ μεγάλη πρόοδο πέρα από το θέμα της παιδικής εργασίας και εδώ συμφωνώ με την προηγούμενη ηλίθεια. πέθαναν 287 εργαζόμενοι σε αυτό το κλειστοφοντερικό εργοστάσιο στο Πακιστάν. Τέταρτο, πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Να με συγχωρείτε, τελειώνω. Θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Όταν ε, ότι δεν ενδιαφέρεται ο καταναλωτή, εμεί πρέπει να το δούμε αντίστροφα το πρόβλημα και να ζητήσουμε από τι μεγάλε επιχειρήσει. Αν ήξερε ο καταναλωτή ε, ότι έχετε υπεργολαβία στην Κίνα, είναι «Ε, όχι, όχι. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λοιπόν για τη διαφάνεια, για το από πού έρχονται τα προϊόντα. Αυτό είναι θεμελιώδη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στην ε, τρίτη εμπειρογνώμονα, την κυρία Σουζάν Στόρμερ. Είστε αντιπρόεδρος ε, του Global TBL Management, μιας ε, φαρμακοβιομηχανίας στη Δανία, Novo Nordisk και είναι υποδειγματική επιχείρηση από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό το σκανδιναμικό μοντέλο σε ό,τι αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Thank you. I will do what I can. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ιδιαίτερα τον κύριο Χάουερτ. Η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε ήταν περίπου 10 χρόνια πριν, εδώ στις Βρυξέλλες, όταν η Novo Nordisk μαζί με εμένα βρεθήκαμε εδώ για να παραλάβουμε ένα βραβείο για την καλύτερη υποβολή εκθέσεων για την βιωσιμότητα. Πιστεύω πως όπως και η συνάδελφοί μου έχει... έχουμε δει μεγάλη πρόοδο και με μεγάλη μου χαρά λοιπόν ήρθε εδώ να σας μιλήσω εκ μέρους της εταιρείας των παρόμοιων εταιριών αλλά και ως πολίτης που ενδιαφέρεται για το ζήτημα αυτό. Καταρχάς ε, θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και να τους ε, συγχαρώ για την... και να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και θα ήθελα σε κάποιο σημείο να συζητήσουμε και το εταιρικό σκέλος. Διότι παρατηρούμε μία διαφορά ανάμεσα στην οικονομική και την κοινωνική διάσταση. Δηλαδή, της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Και αυτό πιστεύω ότι μας κάνει να χάνουμε το στόχο. Εμείς από την άποψη της ε, την εταιρική μας άποψη της αγοράς πιστεύουμε ότι μια υγιής οικονομία είναι η βάση για μια εται... Ε, υγιή επιχείρηση. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε πως μπορούμε να συνεισφέρουμε στην ευημερία της κοινωνίας Και επίσης έχουμε επίγνωση ότι ο ρόλος μας είναι να υπηρετούμε την κοινωνία. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τώρα έχουμε αρχίσει και χάνουμε την γενική ε, εικόνα, ότι δηλαδή το κλειδί της μιας επιχείρησης είναι να υπηρετεί την κοινωνία. Με την ε, κοινωνική εταιρική ευθύνη η κοινωνική εταιρική ευθύνη για μένα έχει τρεις πτυχές. Υπεύθυνη συμπεριφορά και αυτό μπορούμε να το κωδικοποιήσουμε σε κανονισμούς, σε νομοθεσίες. Έχουμε κατευθυντήριες γραμμές. Μπορούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο αναμενόμενης συμπεριφοράς. Το επόμενο επίπεδο είναι πώς μπορεί μια επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική. και πώς μπορούμε να χτίσουμε πάνω στις ε, αξίες. Υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο το οποίο ίσως δεν έχει αναλυθεί εκτενώς ακόμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς θα επιθυμούσαμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με άλλους εταίρους στην αντιμετώπιση του, δηλαδή η, συστημική, η θεμελιώδηση συστημική αλλαγή που χρειάζεται ιδιαίτερα στις καινοτομίες πραγματικά χρειαζόμαστε ενάβσματα από πολλές κατευθύνσεις που θα αποτελέσουν πρόκληση για δημιουργία συστημικών αλλαγών. Πρέπει δηλαδή να επιλέξουμε να δούμε την Ευρώπη ως ε, έναν αδύναμο ασθενή ή ως ένα νέο δυνατό μέλος της κοινωνίας. Στόχος μας είναι βέβαια να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά αυτό που θα θέλαμε επίσης είναι να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος και να εργαστούμε εκεί. Και με βάση την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής νομίζω πως αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Να δούμε δηλαδή ποια είναι η ρίζα του προβλήματος και τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις γι' αυτό. Να σας υπενθυμίσω κάτι που αναφέρεται ως το όριο απόδοσης. Υπάρχουν λίγες εταιρείες οι οποίες ελέγχουν το 73% του ΑΕΠ και απασχολούν το 8% του εργατικού δυναμικού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε στο πλευρό μας αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί πραγματικά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η Novo Nordisk, ε, βασισμένη σε αναλύσεις, είναι η πιο σημαντική εταιρεία στη, στη Σκανδιναβία. Και ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι να υπηρετούμε την κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Διαπιστώνουμε ότι όσον αφορά τον ορισμό υπάρχει συμφωνία ακούγοντάς σας, αυτό διαπιστώνουμε. Ο κατάλογος των ομιλητών ε, Νάντια. Η Νάντια Χίρς. Καταρχήν σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τις ομιλήτριες για την παρουσίασή σας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το θέμα. Είναι ένα τομέα που φυσικά μπορεί να μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο. Είμαι την προηγούμενη εβδομάδα στην Αμερική, στις Ηνωμένε Πολιτείε και συνάντησα και μη κυβερνητικού οργανισμούς αλλά και ενώσεις επιχειρήσεων με τους οποίους ε, συνομίλησα και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση αυτής της εταιρική ευθύνης ε, από μέρους των Αμερικανών ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφώς και υπάρχει πολλές φορές σε μεγάλες εταιρείες μία κατεύθυνση, ένας προσανατολισμός προς την κοινωνική ευθύνη και αυτό φαίνεται και στη στρατηγική τους και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα κέρδος, ένα όφελος για τις επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται. Και από τη στιγμή βεβαίω που η κατάσταση είναι ωφέλιμη και χρήσιμη για όλους, είναι μια win-win κατάσταση, τότε βεβαίως μακροπρόθεσμα μπορούμε να θέσουμε στόχους και να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον είναι βεβαίως ε, το θέμα της παιδικής εργασίας για μένα πέρα από το θέμα της ε, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης υπάρχει και ένα θέμα ίχνη λασιμότητας. Ε, από πού προέρχονται τα προϊόντα και πώς έχουν κατασκευαστεί, βεβαίως. μπορεί να έχουμε διαφορετική προσέγγιση και κατανόηση κάποιων θεμάτων, αλλά αυτό είναι και θα έπρεπε να είναι μια κοινή βάση. Επίσης, πώς παράγονται και πώς επιτόπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείε εκεί που γίνεται η παραγωγή, έτσι ώστε να έχουν μια θετική δράση σε τοπικό επίπεδο, στην κοινότητα, στο Δήμο, να μπορέσει να υποφεληθεί η κοινότητα, η περιοχή από την δραστηριότητα μιας εταιρείας. Και με αυτόν τον τρόπο όντως θα είναι χρήσιμη και ωφέλιμη για όλα τα μέρη η δραστηριότητα μιας εταιρείας. Η σύγκριση λοιπόν με τις Ηνωμένε Πολιτείε και με την Ευρώπη, εγώ μπορώ να συγκρίνω πολλές φορές με τις γερμανικές εταιρείες, πολλές φορές είναι πολύ πιο επιφυλακτικές οι ευρωπαϊκές εταιρείες και έχουμε την εντύπωση ότι κινδυνεύουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να υποχωρήσουν, να μοιραστούν κάποια από τα κέρδη τους. Θα πρέπει όμως πραγματικά να πάψουν να δικαιολογούνται οι επιχειρήσεις όταν θέλουν να έχουν μια θετική δράση, να κάνουν κάτι καλό μια άλλη συνειδητοποίηση χρειάζεται. Έτσι λοιπόν θεωρώ πραγματικά ότι μπορεί να είναι θετικό να στηρίξουμε, να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις έτσι ώστε να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και ενδεχομένως αυτό θα ήταν σίγουρα πολύ πιο χρήσιμο από το να θέσουμε δεσμευτικά κριτήρια τα οποία δεν μπορεί παρά να είναι τελείως διαφορετικά από τον ένα τομέα και από τον ένα κλάδο στον άλλο. Αυτό νομίζω όμως θα το συζητήσουμε περισσότερο όταν προχωρήσει η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φίλιπ Μπουλόν έχει το λόγο, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω έπρεπε να το είχα κάνει όταν πήρε το λόγο εισηγητής, ότι μία ακρόαση έχει νόημα αν μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις στους ε, εμπειρογνώμονες έτσι ώστε να μας ενημερώσουν για θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Αν έχετε λοιπόν φίλοι, ερωτήσεις ε, μπορείτε να τις κάνετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα μεταφέρω υπομορφή ερωτήσεων τις παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Για να σας υπακούσω. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει ένας κοινωνικός και οικονομικός ρόλος για τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να έχουν αυτήν την κοινωνική ευθύνη και θεωρώ ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ αυτών των δύο πτυχών της εταιρικής δραστηριότητας. Ο κύριος Χάουιτ έδωσε κάποιες προθεσμίες όσον αφορά την διαδικασία αυτή της κοινωνικής ευθύνης. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν βεβαίως και αντιμετωπίζουν προβλήματα διακυβέρνησης και σαφώς και θα πρέπει όλα οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλοι αυτοί που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους στόχους αυτών των επιχειρήσεων που έχουν ε, ευαισθησίες δεοντολογικές, περιβαλλοντολογικές, διακυβέρνησης και κοινωνικής ευθύνης. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Όσον αφορά τα θέματα υπεργολαβίας, τα θέματα μεγέθους. Βεβαίως, το θέμα της κοινωνικής δράσης αυτών των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι τελείως διαφορετικό ανάλογα με τους διάφορους τομείς. Όσον αφορά την κοινωνική επιχείρηση, θα πρέπει εδώ να δούμε ποιες είναι αυτές οι εταιρείε που επενδύουν στον κοινωνικό τομέα. Γιατί κάνουμε τέτοιες διακρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν αυτήν την καθαρά κοινωνική ευθύνη, αυτών που επενδύουν σε τομείς όπως το περιβάλλον ή η κοινωνική πολιτική και των επιχειρήσεων που βεβαίως έχουν σαν κύριο σκοπό το κέρδος, οι οποίες όμως έχουν μία πρακτική στον τομέα του περιβάλλοντος και στον κοινωνικό τομέα παραδειγματική. Γιατί λοιπόν αποκλείουμε ε, αυτών των ε, τομέων όλες αυτές τις εταιρείε. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι δυνατότητες έχουμε να παρακολουθήσουμε αυτές τις κοινωνικές βαθμολογίες, γιατί είναι αρκετά εύκολο να μετρήσει κανείς αυτά τα ε, κριτήρια. Είναι πολύ πιο δύσκολο να μετρήσει κανείς τα κοινωνικά κριτήρια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά εγώ τουλάχιστον προσπαθώ εδώ και αρκετό καιρό να δημιουργήσω ένα σύστημα κοινωνικής βαθμολογίας. Ένας τρόπος δηλαδή να αναλύσει κανείς αυτές τις κοινωνικές εταιρείες, όποιος και να είναι ο τρόπος, αν θέλετε, που είναι κοινωνικές, μπορεί να μην είναι καθαρά εταιρείε που επενδύνουν στο κοινωνικό τομέα, αλλά που έχουν μια κοινωνική δράση παραδειγματική. Θα ήθελα λοιπόν να επιβληθεί αυτή η κοινωνική βαθμολογία και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Πώς θα μπορούσαμε με έναν τρόπο συνεκτικό, με περισσότερη συνοχή δηλαδή, να αντιμετωπίσουμε την ε, κοινωνική αυτή δράση και να τη βαθμολογήσουμε. Να την αξιολογήσουμε με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο ευανάγνωστο για τους επενδυτές οι οποίοι θα ήθελαν να επενδύσουν είτε στις κοινωνικές ε, κοινοφελείς εταιρείες είτε σε εταιρείες με κοινωνική εταιρική ευθύνη. Με αυτό τον τρόπο θα είναι πολύ πιο εύκολο και διαφανές να αξιολογήσει κανείς ε, τη δράση των εταιριών αυτών στον τομέα τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντολογικό. Δεν ξέρω αν ε, συμφωνείτε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει καταρχήν σε προαιρετική βάση, δίνοντας κίνητρα, όχι δηλαδή με δεσμευτικό τρόπο, με έναν τρόπο που θα προσελκύσει τους επενδυτές, ελκυστικό για τους καταναλωτές, αλλά και τις δημόσιες αρχές. Αν δηλαδή υπήρχε μία ρήτρα ε, για τις κρατικές αρχές, για τις δημόσιες αρχές, αλλά και σε όλους τους διαγωνισμούς, παραδείγματος χάρη, είτε τις κρατικές προμήθειες, αν υπήρχε μια κοινωνική ρήτρα που θα βασιζόταν σε αυτή την κοινωνική βαθμολογία, θα μπορούσαμε ενδεχομένω με προαιρετικό τρόπο να προσελκύσουμε επενδύσεις προς αυτό το τομέα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά θα πρέπει να βρούμε τρόπους να συνδυάσουμε τον οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους προσκεκλημένους. Ε, είπαν οι προσκεκλημένοι ότι ίσως θα έπρεπε να βγάλουμε το πληθυντικό. Ε, εγώ όμως ε, θα έλεγα πως θα έπρεπε να μιλάμε και για οικολογική και κοινωνική εταιρική ευθύνη. Επίσης, άκουσα έναν ορισμό, νέο ορισμό για την εταιρική κοινωνική ευθύνη που με βρίσκει σύμφωνη, αλλά θα ήθελα να μου πείτε όλες ε, οι επιχειρήσεις, όλες τις επιχειρήσεις αφορά αυτό το θέμα, τι κάνουμε με τις ε, κοπερατίβες, ε, με τις ενώσεις, με τις επιχειρήσεις ελασφάλισης και εκεί υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δομές παραγωγής. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της υγείας, νομίζω ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό. Είχαμε πολλές συζητήσει στη Γαλλία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είδαμε το θέμα του αμοιάντου, και επειδή επιλέγουν κάποια συγκεκριμένα υλικά μόνος έχουμε πολλούς καρκίνους. Επίσης ε, είχαμε και άλλα ε, σκάνδαλα. Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε με αυτά τα κριτήρια της δημόσιας υγείας, του οβεσμού της υγείας, θα συμπεριλαμβάνουμε και επίσης αυτά τα κριτήρια μπορούν να έρθουν εκ των υστέρων, δηλαδή κάνει μία επιχείρηση, μία επιλογή, έχει κάποιους στόχους και εξετάζουμε τον τρόπο παραγωγής και εκεί βάζουμε κοινωνικο-οικολογικά κριτήρια ή αναρωτιόμαστε ποιος είναι και ο ίδιος ο στόχος της επιχείρησης, δηλαδή μια επιχείρηση που παράγει υλικά που προκαλούν θανάτους. Τι γίνεται εκεί, φύγεται η επιχείρηση αυτή περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του τρόπου δράσης της. Και το θέμα των δημοσίων προμηθειών για μένα είναι κάτι σημαντικό θα μπορούσαμε να μιλάμε παραδείγματο χάρη για κινητήρε δυνάμεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν ε, αυτά τα κοινωνικά και οικολογικά κροτήρια. Και τελευταίο σημείο αναρωτιέμαι και σας ε, ρωτώ για το σύνδεσμο που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε από τη στιγμή που θα αποφασίσουμε ότι έχουμε και άλλα κριτήρια Δηλαδή, πέρα από το ότι πρέπει να έχουμε οικονομικά κριτήρια και πώς συνδέουμε αυτό το θέμα των κριτηρίων και της κοινωνικής και ε, οικολογικής ευθύνης με τα κριτήρια, ε, τα οικονομικά δηλαδή και το ΑΕΠ ε, δεν είναι κάτι που το ξεχνάμε. Θα πρέπει να το συνδέσουμε και εκεί και να έχουμε και κριτήρια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που συνδέονται με το επίπεδο το εθνικό και το διεθνές και να έχουμε και άλλα κριτήρια πέρα από το ΑΕΠ. Ευχαριστώ. Πριν να ξαναδώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, θέλω και εγώ να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Κυρία Βραμσκή, είπατε ότι ίσως θα έπρεπε να θέσουμε το θέμα της πρόσβασης ε, στην δικαιοσύνη και ότι λυπόσασταν δεν αναφερόταν κάτι τέτοιο στο κειμένο της Κομισιόν. Αναφερόμενοι σε αυτό το θέμα, τι σκέφτεστε, τις συλλογικέ αγωγές, ε, είχετε κάτι άλλο Επίσης αναφερθήκατε στο θέμα του ορισμού και είπατε ότι χαίρεστε που υπάρχει προσέγγιση με τους ορισμούς των ΗΕ και το ΕΣΑ και τώρα αυτό αρκεί, πρέπει να μείνουμε εκεί ή θα πρέπει να ασκήσει και άλλη πίεση το Κοινοβούλιο για να πάμε πιο μακριά. Τρίτη ερώτηση. Κάποιο ε, εξημώνα ή ε, κυρία Ρώσκη πάλι είπε ότι χαίρεται πολύ που υπάρχει, μάλλον να υπάρχει πιο στενή σχέση μεταξύ εταιρικών, ε, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κυβέρνηση των επιχειρήσεων και εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτά τα θέματα παράλληλα τα βλέπουμε και στο πλαίσιο της Επιτροπής, όμως νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να ελοπίσουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η διαχείριση των επιχειρήσεων, η διακυβέρνηση των επιχειρήσεων και η αμφισημία που υπάρχει για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ότι δεν ε, πρέπει να υπάρχει σκληρή προσέγγιση, αλλά τελικά δεν ε, αλλάζει ουσιαστικά η προσέγγιση των επιχειρήσεων ε, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ή την πρόσληψη του προσωπικού. Μήπως εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε ένα χρήσιμο μοχλό. Και για το θέμα του υποχρεωτικού ή μη χαρακτήρα. Εγώ δεν την κατανοώ αυτή τη συζήτηση, ειλικρινά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δική μας μέχρι αποδείξεως του Ντίου. Και έτσι λοιπόν έχουμε ε, τον απόλυτο κανόνα του ανεξάρτητου και θεμετού ανταγωνισμού. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να μιλήσουμε και για το ε, θέση κριτηρίων. Και πρέπει να θέσουμε κριτήρια και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Δηλαδή γιατί να μην ε, καταστήσουμε υποχρεωτικά αυτά τα κριτήρια σύγκριση σε κάτι που λειτουργεί. Και ε, γιατί ε, να μην έχουμε τις ίδιες συνθήκες για όλους. Τώρα σε σχέση με το είπε ο κύριος Χάουιτ στην αρχή. Είπε ότι ήταν αρμόδιος για τις διεθνείς συμφωνίες και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Εσείς πιστεύετε ότι ε, ο τρόπος που συμπεριλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, το σεβασμό των αρχών σε αυτές τις συμφωνίες θα πρέπει να συμπεριλάβει και την εταιρική κοινωνική ευθύνη και κυρίως όταν μιλάμε για επενδύσεις σε τρίτες χώρες. Και μία μαρτυρία να σας πω την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στη Λιέγη με κάποιους φίλους ε, στην έδρα της ArcelorMittal και μπορώ να σας πω ότι όταν είμαστε εκεί επί τόπου, σε ένα τέτοιο μέρος, ε, βλέπουμε ποια είναι τα όρια της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης γιατί είμαι σίγουρη ότι η ArcelorMittal ε, μπορεί να πει στην ανακοίνωσή τη ότι εφαρμόζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη εδώ και εκεί, αλλά η πραγματικότητα είναι μια καταστροφή και εμεί την παρατηρήσαμε, την είδαμε. Και αυτά που είδαμε και στη Λέγη με κάνουν να σκέφτομαι ότι μπορούμε να σημειώσουμε και περαιτέρω πρόοδο. Αυτέ τι ερωτήσεις θέλω να σα θέσω εγώ. Κύριε Σιγητά, εσεί θέλετε το λόγο για να θέσετε ερωτήσει στου εμπειρογνώμονε. I'll be very quick, I want... Θα είμαι σύντομο. Αυτό το ζήτημα της ε, ύφεση και το αν η εταιρική κοινωνική ευθύνη θα επιζήσει και θα ξεπεράσει από αυτή την ύφεση, θα μπορούσατε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ποιος είναι ο ρόλος που θέλετε να παίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει την, ε, τον οργανισμό σας σε αυτόν τον τομέα πολιτικής και επίσης αυτή η επιχειρηματική πλευρά της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, οι αξίες που είναι, οι από κοινού αξίες είναι ένα θέμα που συζητείται συχνά. Τι μπορείτε να μας πείτε πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Θα ακούσουμε λοιπόν τους προσκεκλημένους ε, αντίστροφα σε σχέση με τη σειρά που μίλησαν. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Στόρμερ. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα έχετε περισσότερο χρόνο. Πέντε λεπτά δυστυχώς πρέπει να σας δώσω και τώρα. Ξεκινήστε. Thank you very... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω πως... Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως ε, πυροδότησε έντονες ε, συζητήσεις με όσα είπα. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει πυροδοτήσει ανταγωνισμό. Όμως, οι από αξίες για εμάς σημαίνουν το εξή ότι σκεφτόμαστε πολύ καλά τις επιπτώσεις που έχουν οι πράξεις μας σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Και έχοντας γι' αυτό, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία, και δράσεις οι οποίες θα φέρουν την ε, μεγαλύτερη αξία. Επίσης, κάτι που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον όταν γίνεται λόγος για την εταιρική διακυβέρνηση, και συμμερίζομαι τις παρατηρήσεις της Γερμανίδας ε, Ευρωβουλευτή για τις ε, εταιρείε οι οποίες κάνουν το πράσινο λεγόμενο ξέπλυμα. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπορείς να, δεν μπορείς να κάνεις κάτι και να φαίνεται κάτι διαφορετικό στα χαρτιά. Και πιστεύω ότι αυτό που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν ε, είπα ότι θα μπορούμε να φτάσουμε στην λύση, στη ρίζα του προβλήματος, είναι το πώς θα γίνουν οι εταιρείε περισσότερο βιώσιμες. Και εδώ έρχομαι στην εταιρική βιωσιμότητα. Αυτό έχει να κάνει με το πώς μια εταιρεία θα συνεχίσει να υφίσταται, θα συνεχίσει να λειτουργεί ομαλά και αυτό είναι κάτι, η εταιρική δηλαδή βιωσιμότητα είναι κάτι που πρέπει να εισαχθεί στην εταιρική διακυβέρνηση. Και για να είμαι ειλικρινής, πάρα πολλές εταιρείες, ακόμα και μικρές εταιρείες, μπορούν να υποφεληθούν και να, από αυτό και να το εισαγάγουν. Δεν είναι κάτι που αντέχει, που μπορούν να το κάνουν μόνο οι μεγάλες εταιρείες. Σύμφωνα με πρόσφατα πειράματα που έγιναν με επενδυτές οι οποίοι ζήτησαν πληροφορίες από εταιρείε οικονομικές και μετά κοινωνικές, αυτό που είδαμε ήταν ότι όταν οι επενδυτές έλαβαν τις, ε, και τις δύο αυτές πληροφορίες ταυτόχρονα, είχαν την τάση να τις αξιολογήσουν πιο ολοκληρωμένα και αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιώ για να τονίσω την σημασία της εισαγωγής αυτών των στοιχείων στις, ε, στις υποβολές εκθέσεων. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα από πλευράς επενδυτών και πιστεύω πως ε, τα ίδια επιχειρήματα θα μπορούσαν να ισχύσουν και για άλλους ενδιαφερόμενους όσον αφορά την αξιολόγηση των εταιριών. Αυτά προς το παρόν. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου. Θα σε ευχαριστώ. Ο Πατρίκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στην εταιρεία Μιτάλ. Έχετε δίκιο και γι' αυτό και θεωρούμε ότι χρειάζεται πλαίσιο για να είμαστε σίγουροι ότι για κάθε περίπτωση υπάρχει και μία απάντηση. Υπάρχει και μία άλλη εταιρεία, βρετανική, που όπως ξέρετε αποτελεί την έμπνευση για το βιβλίο της Κόπολης, δεν αναφέρω ποια εταιρεία είναι. Πρόκειται για μία ιστορία μίας περιοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο με πολλά κοινωνικά προβλήματα και αναφέρεται στην περιοχή αυτή όπου ένα μικρό μπακαλικάκι έγινε μεγάλο σούπερ μάρκετ, υπερκατάστημα και από την άλλη πλευρά της αλυσίδας βεβαίως υπάρχει παραβίαση όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέχρι το Μπαγκλαντές. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μία βάση, ένα κατόφλι όπως είπε και η Επιτροπή. Το κατόφλι αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλους και να μην μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Και μία εταιρεία μπορεί να αναφέρεται στην κοινωνική εταιρική ευθύνη. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι τηρούν και σέβονται όλα αυτά τα κριτήρια. Γι' αυτό και πιστεύω ότι για κάθε μέγεθος και ε, τύπο εταιρείας θα πρέπει τα ίδια κριτήρια να ισχύουν. Η κοινωνική ευθύνη δεν είναι κάτι που σε καμία περίπτωση μπορεί να παραμείνει. Είναι κάτι που θα έλεγα σήμερα είναι ξεπερασμένο. Μπορεί κανείς να προσθέσει τον όρο περιβάλλον ή και άλλα χαρακτηριστικά. Και την ίδια ώρα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προσθέσουμε νέα εργαλεία, νέα μέσα. Θα πρέπει αντίθετα να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε στα βαστικά στοιχεία τα στοιχεία αυτά τα οποία μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Επιπλέον, συμφωνώ και με σας, Πρόεδρε, όταν λέτε ότι η κοινωνική εταιρική ευθύνη στις εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης είναι κάτι το πάρα πολύ ουσιαστικό. Ζούμε σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο και οι Ηνωμένε Πολιτείε σαφώς και αποτελούν ένα από τους κύριους συνομιλητές μας. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ήταν ευαισθητοποιημένος σε αυτά τα θέματα, αλλά όχι μόνο και οι Ηνωμένε Πολιτείε ξεκινάει και η ίδια ευαισθητοποίηση στην Κίνα. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η αναφορά να γίνει πλέον μία συνιστόσα όλων των εμπορικών συμφωνιών και συνομιλιών. Και ανησυχώ, ανησυχώ πολύ για διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή την εποχή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας άλλης μεγάλης χώρας. Μας απασχολεί το θέμα αυτό, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Έλλην Μπρούσκη. Σα ε, merci beaucoup. Ε, pour... ευχαριστώ για να απαντήσω για το θέμα της αξιολόγησης, της κοινωνικής αξιολόγησης των εταιριών. Όπως είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαληθεύσουμε ότι πράγματι στο σύνολο της αλυσίδας ότι γίνονται απόλυτα σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό περαιτέρω και να δούμε πώς θα μπορούσε να τεθεί στην πράξη. Από την άλλη όμως το να απαιτούμε μεγαλύτερη διαφάνεια από την πλευρά των εταιριών τελικά θα τους ωφελήσει όλους. Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι ανέφεραν το κόστος ε, για μια υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων. Όμως εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μετρήσουμε και ποιο είναι το κόστος της έλλειψης εμπιστοσύνης από την πλευρά των επενδυτών ή των καταναλωτών στις επιχειρήσεις αυτές. Και τις πληροφορίες τις έχουν οι επιχειρήσεις, απλώς θα έπρεπε να τις διαθέσουν στο σύνολο των ενδιαφερομένων μερών για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προληπτικές στοιχές ε, της εταιρική κοινωνικής ευθύνης, ε, η έννοια της δεούσα επιμέλειας ε, που παρουσιάζεται από τον Τζον Ρέγκη στις κατευθυντήρες γραμμές μας φαίνεται ενδιαφέρουσα. Για, για το εξή. Οι επιχειρήσει θα έπρεπε να εντοπίσουν του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με μεσία-μεση επίπτωση, να προβλέψουν τις αρνητικές ε, επιπτώσεις και αν χρειαστεί να ε, επανορθώσουν. Και ουσιαστικά στα θέματα δημόσιας ε, υγείας θα μπορούσαν να δράσουν σε ένα στάδιο πριν να υπάρξουν οι παραβιάσεις σε ό,τι αφορά το θέμα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και σε σχέση με τις συλλογικέ αγωγές. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει μία από τις λύσεις που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλες, πρέπει να αναρωτηθούμε σχετικά με τα νομικά εμπόδια για τα θύματα των τριών των χωρών, πόσο δύσκολο θα ήταν ε, να έχουν ε, πρόσβαση στα ευρωπαϊκά δικαστηρία άνθρωποι αυτοί και να ενδιαφερθούμε και για το κόστος ε, που θα σημαίνει αυτό για τα θύματα για να προσφύγουν στην Ευρώπη, να καταθέσουν μια αγωγή στην Ευρώπη. Ήδη έχουν γίνει εργασίες στο επίπεδο αυτό και περιμένουμε από την Κομισιόν να δώσει μια συνέχεια σε αυτή τη μελέτη η οποία αφορά το νομικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Δεν σημείωσα άλλες συγκεκριμένες ερωτήσεις. περιμένουμε από την Κομισιόν. Ίσως να δημοσιεύσει την έκθεση αυτή για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τα τέλη του 12, αν είναι δυνατόν. Και να συμμετέχουν και διάφορες γενικές διευθύνσεις στη διαδικασία αυτή, γιατί μέχρι τώρα δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Σας δίνω το λόγο για να ολοκληρώσετε. Μάλιστα. Γνωρίζω ότι ο συνάδελφο τη Γενική Διεύθυνση άκουσε πάρα πολύ προσεκτικά, όπω και όλοι. Δυστυχώ δεν του επέτρεψε ο χρόνο να μιλήσουν, όμω πραγματικά εκτιμούμε την δουλειά του. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ιδιαίτερα στην κυρία Χίου και στον κύριο Μπουλόν ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη, για συνεισφορά του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρειαζόμαστε όσο μεγαλύτερη συνένεση μπορούμε. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι ήσασταν πάρα πολύ εργατικοί προς αυτό το πράγμα. Κυρία Χίους, ε, έγιναν συνομιλίες με, του, με Αμερικανούς συναδέλφους για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αναφέρθηκαν πολλά ζητήματα, αναφέρθηκαν λοιπόν πολλά και αυτό που το ερώτημα που προέκυψε είναι γιατί δεν κάνετε περισσότερα. Πιστεύω πως πρέπει να έχουμε ταπεινοφροσύνη. Το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, δείγμα ήταν παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα όμως δεν είμαστε. Και πραγματικά έχουν γίνει πολύ σωστέ παρατηρήσεις όσον αφορά την παιδική εργασία. Συμφωνώ με εσά ότι δεν είναι τόσο προφανέ όσο θα έπρεπε να είναι. Όλοι μιλούμε για την εκμετάλλευση τη παιδική εργασία και την καταστροφή τη υπόλοιπη ζωή των παιδιών εξαιτία αυτού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, πολλέ εταιρείε να μπορούν να δηλώσουν ότι δεν χρησιμοποιούν παιδική εργασία. υπάρχει μια νέα πρωτοβουλία όσον αφορά τις εθελοντικές ενέργειες και πολλές επιχειρήσεις ήδη έχουν αναλάβει και υιοθετήσει αυτή την πρωτοβουλία. Και όσοι κάνατε λόγο για διαφάνεια, και εσείς κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω πως ε, αυτό είναι μια συνέχεια της ε, δήλωσης του Ρίο Συνήκωση, ότι ο κόσμος προχωρά, ότι έχουν δημιουργηθεί διάφοροι κανονισμοί σε χώρες όπως την Νότια Αφρική και σύντομα στην Ινδία. Πρέπει λοιπόν να διεξάγουμε τη συζήτησή μας εδώ με ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερα όσον αφορά τη Γερμανία. Θα ήθελα να πω για την, στην ε, κυρία Χίρς ότι σχετικά με αυτά που είπε για τις γερμανικές επιχειρήσεις ότι σχεδόν ντρέπονται να πούν ότι έχουν δράση κοινωνική εταιρική ευθύνη, ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη συνεισφορά σα. Σε αυτήν εδώ την Επιτροπή δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά αυτό το ζήτημα, όμως εγώ θέλω να ασχοληθώ με το ζήτημα της διαφάνειας. Κύριε Μπουλόν τώρα, κοινωνικές επιχειρήσεις, fair trade, αμοιβέ δράσεις, όλα αυτά είναι ένα παράδειγμα κοινωνικής εταιρική ευθύνης. Δεν θέλουμε φυσικά να χάσουν αυτές οι εταιρείε το μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά, αλλά θέλουμε να τις οθήσουμε να αναλάβουν εταιρική κοινωνική ευθύνη και να ασχοληθούν με αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τονιστεί η σημασία αυτής της ε, νέας εταιρικής κοινωνικής πρωτοβουλίας. Επίσης, πιστεύω ότι όσον αφορά την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα αρκετά δύσκολο έργο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι έχει γίνει πρόοδος. Αλλά δεν είχαμε την επιτυχία που θέλαμε. Και συμφωνώ με αυτό που είπατε όσον αφορά τις επενδύσεις επίσης. Κύριε Μπένεραπ, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε. Και εδώ θα ήθελα να μιλήσω για τον ορισμό και να απευθυνθώ σε όλους σας. Ακούσαμε τα συνδικάτα, ακούσαμε τις επιχειρήσεις ε, που, και που μας είπαν ότι είναι σύμφωνοι με αυτόν τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την, ε, την επαγγελματική ηθική, την κοινωνική διακυβέρνηση, την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αλλά στην ουσία όλα αυτά που λέμε είναι το ίδιο πράγμα. Και πιστεύω ότι πραγματικά θα γλιτώσουμε πάρα πολύ χρόνο εάν απλά δεχτούμε τον ορισμό τον οποίο διατύπωσε η Επιτροπή στο έγγραφό της. Και πρόεδρε, όσον αφορά αυτό που είπατε, αναφέρθηκε μια, ένα έξυπνο σύνολο στις επιχειρήσεις. Μια μίξη, μια σωστή και έξυπνη μίξη. Και αυτό πιστεύω πως είναι κάτι με το οποίο μπορούν να συμφωνήσουν όλοι και αναφέρθηκε και στο έγγραφο της Επιτροπής. Θα επιθυμούσα το έγγραφό μου εδώ να ασχοληθεί με το ζήτημα της ανάκτησης στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και εδώ θα θέλω να ζητήσω την συνεισφορά όλων εσάς. Πολλές εταιρείες βρίσκονται στο προσκήνιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, περίπου 6.000 εταιρείες παγκοσμίων δημοσιοποιούν στοιχεία για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αλλά στην Ευρώπη έχουμε περίπου 70.000 πολυεθνικές εταιρείες και υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Επίσης, ακούστηκαν οι από κοινού κοινέ αξίες. Τις ανέφερε ο συνάδελφος οι εξή αυτέ πρέπει να είναι από κοινού για όλους τους ε, ενδιαφερόμενους. Πάντως σε, σε γραμμέ γενικές γραμμές ε, απόλαυσα πάρα πολύ αυτήν την συζήτηση και είμαι σίγουρο ότι, ότι από αυτήν την ακρόαση θα δημιουργηθεί μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζητήσει και πραγματικά ελπίζω να ε, επιτύχουμε συνένεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Συμφωνώ μαζί σας και εγώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, τρεις προσκεκλημένους για τις παρουσιάσεις τους για την Επιτροπή μας. Είναι μια μεγάλη και σημαντική συνεισφορά. Θα βασιστούμε σε αυτά που μας είπατε και θα τα ενσωματώσουμε στην ε, έκθεση του Richard Howitt. Τώρα, όσον αφορά τον ορισμό, δεν διαφώνησα, απλώς ε, έκανα μία ερώτηση. Φαίνεται ότι απαντήσατε. Σημειώνω. Εγώ δεν είμαι τόσο ειδήμων για το θέμα αυτό και απλώς ρώτησα, ρώτησα αν μας αρκεί αυτό που συμβαίνει ή αν ε, θέλουμε κάτι παραπάνω. Αν όλοι είναι ικανοποιημένοι από τον ορισμό αυτό, μου αρκεί και εμένα. Ευχαριστώ και την Επιτροπή και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στις ημερομηνίες. Στις 19 Νοεμβρίου θα υποβάλλετε το σχέδιο του κειμένου σας. Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου μπορούν να υποβληθούν τροπολογίες οι οποίες θα εξεταστούν στις 6 Δεκεμβρίου και θα υιοθετηθεί το σχέδιο στις 14 Ιανουαρίου. Πάντα σε διαβούλευση με την Νομική Επιτροπή. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 31. Ο Στίβεν Χιούζ έχει το λόγο. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας όσον αφορά τις απειλές εναντίον της υγείας στο χώρο εργασίας λόγω αμοιάντου. Πρακτικές εξάλληψης του υπάρχοντος αμοιάντου. Ο εισηγητή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, είχα κάνει στην περισμένη συνεδρίαση μια αρκετά εκτεταμένη εισαγωγή και εμπειρογνώμονες σε εκείνη την ακρόαση υποστήριξαν τα κύρια σημεία τα οποία παρουσίασα τώρα. Οι ε, συνάδελφοι έχουν την έκθεση ενωπιών τους. Η προθεσμία για τις τροπολογίες θα είναι 18 Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν, ε, ανυπομονώ να στείλετε τις τροπολογίες σας και να συζητήσω με τους σκιώδεις πέρα από το θέμα αυτό για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συνεννόηση. Να κάνω τώρα ε, κάποια εισαγωγικά σχόλια, κάποιες παρατηρήσεις θα μπορούσα να πω, Πρόεδρε, ότι πριν 30 χρόνια η πρώτη έκθεση που συνέταξε ως νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ε, στο θέμα του ομοιάντου και εγώ είπα ότι δεν θα δέσω υποψηφιότητα του 2014. Έτσι λοιπόν ε, είναι ουσιαστική η έκθεση αυτή και ελπίζω να έχει καλά αποτελέσματα. Αλλά πολλά έχουν γίνει αυτά τα τελευταία 30 χρόνια. Φυσικά δεν έχουμε πλήρη απαγόρευση στην αγορά και στη χρήση του αμοιάντου, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε εκατομμύρια τόνους αμοιάντου που είναι κλειδωμένες στι υποδομέ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και στις μεταφορές κυρίως στους δρόμου και στα πλοία. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να βρίσκουν μπροστά του αμοιάντου τα επόμενα έτη δύο σημαντικά θέματα για τον Αμίαντο. Καταρχήν, έχουμε μια πολύ μεγάλη ε, περίοδο λανθάνουσα ε, και μπορεί κάποιος που έχει εκτεθεί να μην ε, πεθάνει για 30 ή 40 χρόνια ε, ως αποτέλεσμα της έκθεσης. Είχαμε ένα μέλος εδώ, τον Άλεξ Φόκνερ, ο οποίος εργαζόταν στα ναυπηγεία στα Φόκλαντ και πέθανε τον Αύγουστο, κατέληξε τον Αύγουστο. Και κάτι για... αυτό είναι η ενθάνουσα περίοδος, ε, το ένα σημείο. Επίσης, δεύτερον, δεν υπάρχει κατόφλι για την έκθεση στον αμίαντο, κάτω από το οποίο ένας πολίτης ή ένας ε, εργαζόμενος θεωρείται ότι δεν κινδυνεύει από έκθεση στον αμίαντο. Αυτό πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Επίσης, ε, έχουμε δύο, παρά, δύο, μία παράλληλες εξελίξεις που δημιουργούν πρόβλημα. Ότι τα υλικά που περιέχουν αμύαντο έχουν ε, κύκλο ζωή 30-60 έτη. Και αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα κτίρια που περιέχουν αμύαντο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, είτε να ανακαινιστούν είτε να κατεδαφιστούν. Και αυτό σημαίνει ότι θα εκτίθενται οι εργαζόμενοι στον αμύαντο. Αλλά όσο ε, περισσότερο, τόσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος αυτή, τόσο λιγότερο είναι εξοικειωμένοι οι εργαζόμενοι με το πρόβλημα. Αυτή είναι η πρόσθετη δυσκολία. Τώρα να αναφέρω τα κυρία στοιχεία της έκθεσης. Ελπίζω όλοι να είχατε την ευκαιρία να τη διαβάσετε και σίγουρα οι σκιώδεις θα είχαν την ευκαιρία να τη διαβάσουν. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε σοβαρά την ανάγκη για πλήρη έλεγχο και ένα πλήρε μητρό για τα υλικά που περιέχουν αμύαντο στι υποδομέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πολλά έτη οι εταιρείε ε, συστήνουν τα δικά του μητρώα σε σχέση με αυτά τα υλικά, όμω νομίζω ότι πρέπει να το ομαδοποιήσουμε σε εθνικά μητρώα για να ε, δούμε πώ θα οργανώσουμε με τις μελλοντικέ εργασίες ανακαίνησης ε, ή κατεδάφισης. Επίσης, δεσμευτήκαμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια, Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου την ανάγκη για καταγραφή και σύνδεση με αυτό το έργο για να βελτιώσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε και την ασφάλεια ένα άλλο θέμα αφορά την προσόντα και την κατάρτιση και την ε, αδειοδότηση. Έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά ε, την χορηγήση αδειών και τα προσόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει κάποια εναρμόνιση ως ένα βαθμό. Η ε, ανάπτυξη προγραμμάτων απομάκρυνσης είναι ο επόμενο τίτλος στην έκθεση. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση εδώ, κύριε Πρόεδρε. Το πυρήνα αυτή τη έκθεση είναι ότι θα πρέπει να καταρτήσουμε σχέδια για την απομάκρυνση του αμύαντο. Υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει ότι αν έχει σφραγιστεί ε, ο αμύαντο κατάλληλα, καλύτερα είναι να μείνει εκεί που έχει. Θα ήθελα να κάνω αυτή τη συζήτηση εδώ, να δούμε τι πιστεύει η πλειοψηφία. Αλλά ακόμη και αν είναι αλήθεια, να πούμε ότι είναι καλύτερα να αφήσουμε τον αμύαντο εκεί αν είναι ασφαλώ σφραγισμένο και πάλι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα και πάλι πιστεύω ότι το θέμα του έλεγχου και του μητρώου είναι σημαντικό το επόμενο αφορά τα κριτήρια αναγνώρισης ε, των ασθενειών σχετιζόμενων με τον αμύαντο. Έχουμε πάρα πολλέ διαφορέ μεταξύ των εθνικών συστημάτων, των εθνικών προτύπων και διαδικασιών ε, για την αναγνώριση, τον εντοπισμό και την αποζημίωση που θα χορηγείται για τι ασθένειε που σχετίζονται με τον αμύαντο. Πρέπει να το δούμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατόπιν υποστήριξη ομάδων θυμάτων αμοιάντου. Αυτές οι ομάδες θυμάτων αμοιάντου εκπροσωπήθηκαν στην προηγούμενη ακρόση που είχαμε. Κάνουν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για να υποστηρίξουν τα θύματα που έχουν εκτεθεί στον αμοιάντο και τις οικογένειές τους και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν το δίκτυό τους και θα πρότεινα ίσως εδώ θα πρέπει να δώσουμε και κάποια οικονομική στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους. Το τελευταίο τμήμα έχει να κάνει με τις στρατηγικές καθολικής απαγόρευσης του ομοιάντου. Είχαμε μία νίκη πρόσφατα, καθώ κάποια ερωτήματα τέθηκαν και στα Εθνικά Κοινοβουλία και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση του Καναδά απέσυρε μία. Ε, επιδότηση που ήθελε να δώσει στο ορυχείο Τζέφρις. Ε, έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσει στον Καναδά η παραγωγή αμοιάντου κατά πάσα πιθανότητα, όμως συνεχίζεται στη Ρωσία. Και καθώς ε, τις προάλλες ε, ε υπήρξε κάποια αναμετάδοση ε, για μια περίπτωση με μία με χρυσοτήλη, ο πρόεδρος Πουτίν τους ε, συνεχάρει αυτούς τους ε, εργαζομένους και τους ε, συνεχάρει που προωθούν τη χρυσοτήλη στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε εμπορία της χρυσοτήλης πριν 40-50 χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε ευθύνη να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Παραδείγματος χάρη είναι λάθος τα ευρωπαϊκά πλοία ε, να στέλνονται στο Μπαγκλαντές ε, και στην Ινδία και να διαλύονται από παιδιά τα οποία εκτίθενται σε αυτές τις ουσίες. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εγώ συναντήθηκα με, εκπρόσωπο μιας πολυεθνικής ε, στο γραφείο μου και μου είπε, μα αυτό δεν έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή απασχόληση το τι συμβαίνει στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η απάντησή μου ήταν, θα έπρεπε να έχει κάποια σχέση με τη δουλειά μας εδώ και την Επιτροπή Επασχόληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί έχουμε ηθικό καθήκον να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε περαιτέρω θανάτου στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτή είναι μια σύντομη εισαγωγή, Πρόεδρε, για το ποια είναι η συλλογιστική της έκθεσης, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τι απόψεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαχ. Μπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στίβεν Χιούς για αυτή την πολύ τολμηρή και εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Φυσικά φαίνεται ότι έχει εμπειρία, φαίνεται και σε αυτήν την έκθεση και βρήκε τον σωστό τρόπο να παρουσιάσει το θέμα αυτό. Πρόκειται για μια επικίνδυνη ουσία και σαφώς και υπάρχει και πολλής χρόνος μέχρι να παρουσιαστούν τα πρώτα συμπτώματα ε, της ασθένειας. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πολύ περισσότερα θύματα ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από τον αμίαντο. Ακόμα και σε μικρές χώρες Σήμερα υπάρχουν υψηλοί αριθμοί εργαζομένων που καθημερινά συνεχίζουν να είναι σε επαφή με τον αμίαντο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτή η καταγραφή και σε άλλα κράτη από αυτά που υπάρχει σήμερα. Θα ήθελα να πω στον εισηγητή πρώτον το θέμα του screening. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται μια ε, πολύ ακριβής ε, καταμέτρηση των κτηρίων, αλλά όχι μόνο των κτηρίων, να υπάρξει μια υποχρεωτική δεσμευτική καταγραφή έτσι ώστε με μεγάλη διαφάνεια να ξέρουμε πού υπάρχει ακόμα αμύαντος. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεύτερον, το θέμα της κατάρτισης των εργαζομένων, ιδιαίτερα των νέων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η ουσία ή γνωρίζουν πολύ λίγα. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, η ευαισθητοποίηση. Αυτό βεβαίως δεν αρκεί. Χρειάζεται και μια εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπάρχουν κοινά σχέδια δράσης. Αυτά τα σχέδια δράσης πιστεύω θα πρέπει να επιβληθούν σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως παραδείγματο χάνει στην Πολωνία. Ξέρετε ότι η Πολωνία εδώ αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με πολύ πρωτοποριακό τρόπο. Πιστεύω θα πρέπει εδώ να χρησιμοποιηθεί αυτό σαν βέλτιστη πρακτική και βεβαίως να υπάρξει χρηματοδότηση η οποία θα επιτρέψει αυτά τα σχέδια δράσης να υλοποιηθούν. Υποστηρίζω λοιπόν την έκθεση και τις προτάσεις ε, του κυρίου Χιούς και πιστεύω ότι θα πρέπει εδώ να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και απαραίτητα να υπάρξει εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσβλέπω στην μελλοντική συνεργασία με τον εισηγητή. Η Μάριον Χάρκιν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω εκ μέλου του συναδέλφου που δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ σήμερα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Χιούς για την λεπτομερέστατη, το λεπτομερέστατο σχέδιο έκθεσης προτείνει ε, αρκετά καλές λύσεις για το πώ θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του αμοιάντου. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν οι απαντήσεις, διότι όσοι εργάζονται σε περιοχές με αμοιάντο διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο υγείας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ρύθμιση των, ε, του, επιπέδων αμοιάντου είναι ικανοποιητική. Η κατεδάφιση των κτηρίων με αμίαντο ρυθμίζεται πολύ αυστηρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αφαίρεση του αμμιάντου απαιτεί πρώτερη συνένεση και έγκριση. Υπάρχουν βέβαια ορισμένε αναφορές για ε, ανθρώπους που εκτέθηκαν σε επίπεδα αμμιάντου σε κτίρια που περιείχαν αμμίαντο κατά τη διάρκεια κατεδαφίστεων και είναι δεν υπάρχει μητρό των ε, εκτεθειμένων ανθρώπων στον αμίαντο και γι' αυτό και δεν μπορεί να γίνει σωστά η ιατρική παρακολούθησή τους. σε πολλέ περιπτώσει, σε πολλά ιατρικά κέντρα, οι γιατροί δεν είναι επαρκώ ενημερωμένοι και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την, ε, αστε, τις ασθένειες που έχουν προκληθεί από αμίαντο. Οι εξετάσεις όμως ε, αυτές για να εντοπιστεί αμύαντος μπορούν να γίνουν μόνο από εξειδικευμένους ιατρούς. Η συναδελφός μου θα καταθέσει τις δικές της τροπολογίες και ελπίζει σε μια επικοδομητική συνεργασία με, με τον εισηγητή. Καρή Μαντέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πρότασή του. Σαν εισηγήτρια για την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανείς ε, τους ε, αριθμούς, τα στοιχεία που έχουμε στην Ευρώπη, είναι πραγματικά ανησυχητικά. 112.000 θάνατοι που οφείλονται στον αμίαντο παγκοσμίω. Και 220 καρκίνοι του πνεύματος που έχουν σχέση με τον αμίαντο. 120.000 άνθρωποι συνεχίζουν να εκτίθενται στον αμίαντο, 80.000 νεκροί που οφείλονται σε ασθένειες που έχουν κάποια σχέση με τον αμίαντο. Πρόκειται για επαγγελματικές ασθένειες και όλα αυτά θα πρέπει πραγματικά να προσθεθούν στην έκθεση αυτή. Θα ήθελα επίσης να πω ότι συνεχίζει να υπάρχει αμίαντος όχι μόνο στα κτίρια, αλλά και στα πλοία. Πρόκειται για μία το οποίο πολλές φορές δεν αναγνωρίζεται. Υπάρχει όμως σε πολλά αντικείμενα τα οποία δεν είναι ακόμα καταχωρημένα. Και κάτι άλλο που πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσει η έκθεση αυτή είναι το θέμα της ευθύνης, ε, ποινική ευθύνης ε, μη του εργοδότη. Υπάρχουν κράτη που ήδη έχουν ε, επιληφθεί του θέματος αυτού και μπορεί κανείς να πει ότι εμείς σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ίσως να κάνουμε ένα βήμα έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση να προσφύγουν στα δικαστήρια Είδαμε ότι στην Ιταλία το ποινικό δικαστήριο του Τωρίνο καταδίκασε κάποιες ε, εταιρείες, κάποιες βιομηχανίες. Πιστεύω ότι στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να συμπεριλάβουμε την ε, βούληση της ε, Ευρώπης ότι θα πρέπει να απαγορευθεί ο αμίαντος παντού. Θα κάνω λοιπόν κάποιες ε, τροπολογίες. Πρώτον, όσον αφορά τα εθνικά σχέδια καταχώρησης των ε, κτηρίων που περιέχουν ε, αμίαντο. Επίσης να υπάρξει μία παγκόσμια απαγόρευση για το εμπόριο του αμοιάντου και των προϊόντων που περιέχουν αμοιάντο και ενδεχομένως μπορούμε να συνδυάσουμε κάποιους στόχους όπως αυτούς της απόδοσης της ενέργειας, να υπάρχουν κάποιοι στόχοι και κάποια κριτήρια για την απαγόρευση και την εξάλληψη του αμοιάντου. Πιστεύω επίσης ότι θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε την έρευνα όσον αφορά την αντικατάσταση του αμοιάντου για να αποφύγουμε μελλοντικές καταστροφές. Θα πρέπει, παραδείγματο χάρη, να απαγορευθεί ο άσπρος αμίαντος. Μια ουσία η οποία σήμερα αμφισβητείται, χωρίς να μπορεί κανείς να αποδείξει την επικινδυνότητα αυτής της ουσίας. Επίσης, τα απόβληπα αμοιάντου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κεραμικών. Επίσης, την αντικατάσταση αυτής της ουσίας για κάποιες κατασκευές που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν ε, τσιμέντο. Θα πρέπει επίσης κανείς να είναι εξαιρετικά αυστηρός όσον αφορά την εξάλληψη του αμοιάντου από τα κτίρια τα οποία κατεδαφίζονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, έχουμε ξεπεράσει την ώρα που είχαμε για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στις βιαστικές ενέργειες όταν θα εξάγουμε συμπεράσματα γι' αυτό εδώ το έγγραφο. Συμφωνώ με όσους πρότειναν ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις ασθένειες που σχετίζονται με τον αμίαντο. Υπάρχουν κτίρια με στέγες από αμίαντο σε πολλά μέρη στην Ευρώπη. Έχουμε ζητήσει να αφαιρεθούν αυτές οι στέγες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ξέρω ότι το κόστος τα αφαίρεσης είναι μεγάλο, αλλά πριν από τρία-τέσσερα χρόνια εγώ ο ίδιο ξόδεψα 3-4 χιλιάδε λίρε για να βγάλω, να αφαιρέσω αμύαντο από τη σκεπή του ίδιου μου του σπιτιού. Και ε, ξέρω ότι ειδικά ε, όσοι αγρότε ε, πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αφαιρέσουν τον αμύαντο θα χρεοκοπήσουν σχεδόν. Υπάρχει αυτό το, αυτός ο κίνδυνο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Δύο λεπτά. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλήστε παρακαλώ, θέλετε να μιλήσετε κύριε Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Σε γενικές γραμμές καλωσορίζουμε την έκθεση αυτή, διότι πιστεύουμε ότι περιέχει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες, τις οποίες γνωρίζουμε. Αν μου επιτρέπετε να εκφραστώ ελεύθερα, Νομίζω πως αυτή η έκθεση πραγματικά πατάει όλα τα κατάλληλα κουμπιά. Αλλά δυστυχώς σε αυτή τη χρονική στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να δεσμευτεί για οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε πράξη. Να σας υπενθυμίσω ότι εργαζόμαστε για αυτό το ζήτημα του αμοιάντου. Πριν από 10 περίπου μέρες δημοσιεύσαμε στον ιστότοπό μας έναν οδηγό για τους εργάτες που εργάζονται σε κτίρια που περιέχουν αμοιάντο. και ενημερώσεις για τις ε, ασθένειες που σχετίζονται με το χώρο εργασίας, για τον εντοπισμό ασθενειών που σχετίζονται με τον αμίαντο στο χώρο εργασίας. Αυτό γενικότερα το ζήτημα θα θέλαμε να το δούμε να εξετάζεται υπό το ε, πρίσμα των ασθενειών που σχετίζονται με το χώρο εργασίας. Ελπίζουμε να έχουμε τελειώσει μέχρι το τέλος του μήνα και θα δείτε ότι στις προτάσεις μας θα βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις και πολλές ενδιαφέροντα στοιχεία ε, όσον αφορά τον εντοπισμό ασθενειών που προκαλούνται από αμίαντο. Φυσικά εμείς προτιμούμε να λύσουμε το πρόβλημα των ασθενειών που προκαλούνται από αμίαντο στο χώρο εργασίας μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των ασθενειών στο χώρο εργασία και όχι να δώσουμε μία συγκεκριμένη λύση μόνο για τον αμύαντο ξεχωριστά. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε τη μελλοντική μας στρατηγική. Εγώ θα προσπαθήσω να πιέσω για απαντήσεις και για αντιδράσεις, ιδιαίτερα στο θέμα του αμοιάντου αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να θεσμευτούμε για κάτι παραπάνω. Και χιούς συμπέρασμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν αναμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει κάποια διέσμευση αμέσως τώρα, όμως μπορούμε να το συμπεριλάβουμε ίσως στην έκθεση και να αναπτύξουμε μια στρατηγική. Θα μπορούσαν λοιπόν τότε να δεσμευθούν. Να απαντήσω στον κύριο Μπένιον. Πιστεύω πως αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια νύχτα. Αναφερθεί ε, αναφέρθηκε ένα συνάδελφο στην κατάσταση στην Πολωνία, η οποία δεσμεύτηκε μέχρι το 2032 να έχει εξαλείψει τον αμύαντο από την επικράτειά τη. Και αυτό πιστεύω πω είναι αρκετά ρεαλιστικό όσον αφορά το χρόνο και το, τον όγκο του έργου που πρέπει να γίνει. Όμω πρέπει να διεξαχθεί μια συζήτηση για το αν πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ή όχι. Και πάνω σε αυτό θα αναμείνω τις ε, τροπολογίες ιδιαίτερα από τους κοιότητες εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 18 Νοεμβρίου. Θα τις εξετάσουμε στις 6 Δεκεμβρίου και θα υιοθετηθεί το σχέδιο γνωμοδότησής σας στις 24 Ιανουαρίου. Εάν και εφόσον έχουμε προηγουμένως λάβει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Στο σημείο 32 πρόκειται την ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους, πρόβλεψη και διαχείριση της αναδιάρθρωσης. Είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ μία μελέτη που έχει προετοιμάσει η μονάδα για την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της εξέτασης ενός κειμένου δικού μας. Πριν δώσω το λόγο στην ε, μονάδα αυτή, δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή και κατόπιν στους τέσσερις ειδικούς. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονε και να πω στους συναδέλφου, όπως σας δούμε στο επόμενο σημείο, ότι το έγγραφο αυτό που θα μας παρουσιάσουν θα είναι, τουλάχιστον αυτό ελπίζω εγώ, αυτό που θα πυροδοτήσει την κατανοήσή μας ε, όλων των λεπτομεριών και των ιδιαιτεροτήτων ενός τέτοιου πολύπλοκου θέματος. Εγώ ως εισηγητής θεώρησα ότι έπρεπε να ζητήσω τη βοήθειά του για να μας αποσαφηνίσουν αν υπάρχει πράγματι προσθεμένη αξία και ποιο είναι το κόστος και τα ωφέλη. Και Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ερμηνείες που είναι μακριά από την πραγματικότητα, όμως ε, ε, ούτε εγώ προσωπικά, ούτε κανένας από το προσωπικό στο γραφείο μου δεν είχαμε καμία ε, σχέση. Η ενότητα έκανε την έρευνα αυτή. Εγώ ελπίζω να έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα που θα τα χρησιμοποιήσουμε στο έργο μας. Σας ευχαριστώ και πραγματικά έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να ακούσω τις παρατηρήσεις σας ε, και πολιτική αλλά και προσωπική. Σας ευχαριστώ. Ε, ναι, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάρλα από το Πανεπιστήμιο του Βόρικ. Ναι. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Sorry. Yes, thank you for asking me here to speak today. Uh, my uh, ευχαριστώ πολύ. Το όνομά μου είναι Mark Carley. Κατάλαβα ότι είμαι καθηγητής αν διαβάσω το έγγραφο. Δεν ε, ισχύει όμως αυτό. Εν πάση θα σας μιλήσω για τις δυνατότητες της ε, ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας όσον αφορά την ευρωπαϊκή αναδιάρθρωση και θα βασιστώ βεβαίως στο σχέδιο ε, έκθεσης. Θα παρουσιάσω σύντομα τα συμπεράσματά μου. Πιστεύω ότι στην έκθεση που σας έχει μοιραστεί μπορείτε να δείτε την ουσία αυτών που θα ήθελα να σας παρουσιάσω. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εξετάζω την παρούσα κατάσταση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξετάζοντας ιδιαίτερα την ομοθεσία, τις συλλογικέ συμβάσεις και την ε, παρέμβαση των δημόσιων αρχών, καθώς και την πρακτική των ε, επιχειρήσεων. Τα συμπεράσματά μου είναι ότι η παρούσα κατάσταση στα κρατη σε αυτούς τους τομείς που ασχολείται η αναδιάρθρωση, είναι πολύ διαφορετική υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ε, εμπλεκόμενων ε, μερών όσον αφορά τη διαχείριση, την πρόβλεψη, όπως φαίνεται από το σχέδιο έκθεσης. Όμως αυτές οι πρακτικές, από ό,τι φαίνεται και διαπιστώνεται, δεν ισχύουν σε πολλές επιχειρήσεις και δεν αφορούν πολλούς εργαζόμενους. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης όσον αφορά την φύση των πρακτικών των επιχειρήσεων και ότι σε πολλούς τομείς και σε πολλές επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι φαίνεται να μην υποβάλλονται σε απολύτως κανένα πρότυπο, καμία εγγύηση και ότι αυτό οφείλεται και εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των ε, εργοδοτών. Αυτό ισχύει κυρίως ε, για την ε, πρόβλεψη της αναδιάρθρωσης. Τώρα πάρα πολλές εταιρείε ε, μπορούν να εντοπιστούν, να τις δούμε ως παράδειγμα καλών πρακτικών, όπως και στο ότι παρέχουν πολλές συλλογικές συμβάσεις ή κανονίζουν δημόσιες παρεμβάσεις. Όμως ε, φαίνεται να υπάρχει άνεση κατανομή των καλών πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καμία, ε, για καμία χώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα πραγματικά πλήρε και ολοκληρωμένο πλαίσιο και πολιτικών ε, που να προωθεί το μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό των δεξιατήτων, την έγκαιρη προετοιμασία και την κατάλληλη διαχείριση τη αναδιάρθρωσης και την ελαχιστοποίηση του ιστορικού και εξωτερικού κόστου Τη αναδιάρθρωσης. Εξέτασα τα, τις τάσεις ε, στον τομέα αυτή και ε, είδα ότι χωρίς παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μάλλον θα συνεχιστεί το σημερινό σενάριο. Δεν υπάρχουν σημάδια ότι τα κράτη-μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι κινούνται προς οποιαδήποτε σύγκληση στον τομέα αυτό. Η ένδειξη είναι ότι ορισμένε από τι χώρε που ήδη ρυθμίζουν στοιχεία βαλτιστών πρακτικών μέσω τη νομοθεσία ή των συλλογικών συμβάσεων πηγαίνουν παραπέρα προ την κατεύθυνση αυτή και, οδη... και έτσι υπάρχει μεγάλη απόκληση από αυτού που δεν έχουν νομοθεσία και ρύθμιση στον τομέα αυτό. Σαν ε, αυτό είναι εξαίρεση ε, το ότι πολλά κράτη-μέλη απάντησαν στα αποτελέσματα της κρίσης ε, κατά τα έτη 2008-2010 με ορισμένες δράσεις αναδιάρθρωσης, διαχείρισης της αναδιάρθρωσης ε, όμως σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα μέτρα ήταν προσωρινά και βραχυπρόθεσμα και λίγα προσπάθησαν ε, να πάνε παραπέρα ε, από το να ε, καλύψουν άμεσα προβλήματα, να ανακουφίσουν άμεσα προβλήματα και να προετοιμάσουν κατάλληλα τους εργαζομένους και τις εταιρείες έχοντας εξετάσει τη σημερινή κατάσταση, το επόμενο θέμα που εξέτασα είναι ότι τι θα συνέβαινε με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν υπήρχε δεσμευτική μορφή παρέμβασης. Σίγουρα θα υπήρχε υπήρχε νομοθετική αλλαγή για να εφαρμοστούν οι νέε διατάξει στα κράτη-μέλη, Όλε οι χώρε θα υποχρεούνται να εθίσουν σημαντική νέα νομοθεσία, Κυρίω στον τομέα της πρόβλεψης τη αναδιάρθρωση, όπου γενικά τώρα σιωπάει η νομοθεσία. Στον τομέα της διαχείρισης της αναδιάρθρωσης, ο νομοθετικός αντίκτυπο, θα ήταν μάλλον μικρότερο αλλά ε, και πάλι ουσιαστικός ε, σε πάρα πολλές ε, δυτικές ευρωπαϊκές χώρες γιατί υπάρχει δυνομοθεσία ή συλλογικές συμβάσεις σε αυτόν τον τομέα. Μια πιο μεγάλη αλλαγή θα πετούταν στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με κάποιες λίγες εξαιρέσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Δυτικής Ευρώπης είναι υπεράκτιες περιοχές. Τώρα, κάποιες τομείς, σε κάποιου τομεί και εταιρείε, το αποτέλεσμα τη απαιτούμενη νέα νομοθεσία θα μετραζιόταν γιατί θα καλυπτόταν από συλλογικέ συμβάσει που έχουν να κάνουν με σχετικά ζητήματα. Και επομένω, ε, ίσω ε, θα υπήρξε κάποια εξαίρεση από τι ε, ε προτινόμενε υποχρεώσει εκ του νόμου. Τώρα, ε, κάποιες ε, τέτοιες ε, διαδικασίες ε, για την πρόβλεψη και τη διαχείριση ίσως υπάρχουν στη Γαλλία, όμως έχουμε πιο κοινέ συμφωνίες για να προετοιμαστεί με έναν κατάλληλο τρόπο να αναδιάθρωση και να μειωθεί το κοινωνικό κόστος. Έχουμε και προδραστικές συμφωνίες σε χώρες όπως Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Καταχώρες και Σουηδία φαίνεται ιδιαίτερα πιθανή η υιοθέτηση οποιοδήποτε προτιμόμενη νομοθετική πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ε, προωθούσε τι συλλογικέ συμβάσει για την ε, πρόβλεψη και τη διαχείριση τη ενεδράθρωση, ε, δεδομένου το ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα ήθελαν να έχουν ευελιξία σύμφωνα με την ευελιξία που τους προσφέρει η συμφωνία. Όμω μια τέτοια όθηση μπορεί να έχει αποτελέσματα σε χώρε που ανέφερα ήδη, όπω Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία κτλ., που ήδη έχουν κάποιε σχετικέ τέτοιε συμβάσει. Τώρα, αντίκτυπο τη πρόταση στι δημόσιε αρχέ θα ήταν ε, να του απαιτηθεί να ολοκληρώσουν ε, τη σημερινή ε, σχετικά διαρθρωμένη παρέμβασή του και να διασφαλίσουν ότι καλύπτει μια σειρά συγκεκριμένων τομέων, συντονισμό, υποστήριξη, παρακολούθηση τη πρόβλεψη, περιφερειακέ πρωτοβουλίε και χρηματοδότηση μέτρων απασχολησιμότητα. Αν ε, και τα πλήρη στοιχεία για τι σημερινέ παρεμβάσει, δεν είναι διαθέσιμα, φαίνεται ότι οι περισσότερε χώρε θα έπρεπε να εφαρμόσουν τουλάχιστον κάποιε νέε παρεμβάσει. Έτσι λοιπόν, για να συνοψίσω η κλίμακα και τα αποτελέσματα τη προτινόμενη πρωτοβουλία, ε, θα ήταν πολύ σημαντικά και θα οδηγούσαν σε μεγάλε νομοθετικέ αλλαγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ε, αφορούσαν χιλιάδε εταιρείε. Οι νομοθετικέ αλλαγέ θα ήταν πολύ ευρύτερε από αυτή που απαιτείται από την οδηγία πλαίσιο του 2002 για την ενημέρωση και διαβούλευση που ουσιαστικά ζητούσε πολύ μικρά μέτρα που έπρεπε να ληφθούν στο ιστορικό δίκαιο των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την ε, ανάλυση των γεγονότων, πριν και μετά, εξέτασα και τα επιχειρήματα σε σχέση με το επίπεδο και τη φύση οποιασδήποτε παρέμβαση στην αναδιάρθρωση και τα αποτελέσματα της προηγούμενης δραστηριότητας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετικής και μη νομοθετικής στον τομέα αυτό. Όπως ανέφερα, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις από τις σημερινές τάσεις ότι τα κράτη-μέλη χωρίς ε, όθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να προωθήσουν το ρυθμιστικό τους πλαίσιο στον τομέα αυτό με συνεκτικό τρόπο. Κάποιες χώρες ε, έχουν εισαγάγει σχετική νομοθεσία τα πρόσφατα έτη, όμως η συνολική πρόοδος είναι μικρή, είναι αργή και δεν πρόκειται να πετύχουν το στόχο τους στο εγγύς μέλλον προβλέπω να συνεχίσουν ε, να υπάρχουν τα οικονομικά προβλήματα τα επόμενα έτη και έτσι λοιπόν ε, θα χρειαζόταν ε, πιο διευρυμένη δράση από τη μεμονωμένη δράση των κρατών μελών. Τα άλλα επιχειρήματα που αναφέρω εδώ, βλέπετε, τώρα βιάζομαι γιατί φτάνω στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα των 10 λεπτών, δεν θα τα αναφέρω λοιπόν, αλλά θα Πώ συμπερασματικά σε σχέση με την πιθανή δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση είτε είναι δεσμευτική είτε όχι, εγώ θα τόνιζα ότι ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωση για να προωθηθούν οι πρακτικές σε αυτό το τομέα συγκεκριμένα οι κοινωνικοί εταίροι παρήχαν κάποιους προσανατολισμούς το 2003 στον τομέα αυτό, αλλά δεν φαίνεται να υπήρξε σημαντικός αντίκτυπος στην πράξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολλή δουλειά για να προωθήσει και να διαδώσει τις πρακτικές Επίση για την ε, πρόβλεψη, τη διαχείριση τη αναδιάρθρωση και απασχολησιμότητα, όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την απασχόληση, όμω δεν υπήρξε μια πλήρη απάντηση στι εθνικέ πρακτικέ. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πράγματι να πετύχει πρόοδο στον τομέα αυτό, ίσω θα ήταν καιρό να νομοθετήσει. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη παρουσίαση και θα περάσουμε τώρα στην κυρία Σέμαν, η οποία είναι ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο. Έχετε 10 λεπτά επίσης. Thank you, Chairman, for Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας παρουσιάσω την έρευνα που έχουμε διεξαγάγει που μας ζητήθηκε για την συμβουλευτική σχετικά με τις πληροφορίες. Κοιτάζοντας την αξιολόγηση της ε, προστιθέμενης αξίας των ευρωπαϊκών μέτρων όσον αφορά την ε, συμβουλευτική και την ε, διαδικασία αναδιάρθρωσης, θα δείτε στη διαφάνεια Κοιτάξαμε στην αρχή το συγκείμενο και το συγκείμενο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά το τι αναδιαρθρώνεται και ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε. Και πράγματι, η αναδιάρθρωση είναι μια διαδικασία που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα με ταχύς ρυθμούς και ενδέχεται να οδηγήσει σε έναν μόνιμο κίνδυνο. Και η υλοποίηση αυτών των κινδύνων και των συνεπειών μπορεί να επιφέρει μεγάλες προκλήσεις για όλους τους ε, φορείς, για επιχειρήσεις, για εργάτες, για περιφέρειες. Η αναδιάρθρωση είναι ένα έργο πάρα πολύ περίπλοκο και δύσκολο για να αντιμετωπιστεί από την νομοθεσία και μόνο, είτε την ευρωπαϊκή είτε την εθνική. Και από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, τα μέτρα κυρίως είναι αντιδραστικά παρά δραστικά. Σε, συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένους τομείς, ε, στην ε, συμβουλευτική σχετικά με την πληροφόρηση, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε, το δούμε αυτό και ε, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Παρατηρούμε γενικά μια ασυμμετρία στα μέσα ανάμεσα στους εφορείς, μια συμμετρία στα επίπεδα της ε, λήψης αποφάσεων και μία ανεπάρκεια της ε, ισχύουσας, του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των ε, ευρωπαϊκών μέτρων τώρα. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να δούμε τι έχουμε ποια μέτρα έχουμε στη διάθεσή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να τα αναλύσουμε, καθώς επίσης και να δούμε ποια μέτρα έχουμε στη διάθεσή μας σε εθνικό επίπεδο για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε αν υπάρχει πιθανότητα για να ε, υπάρξει προστιθέμενη αξία, επιπλέον προστιθέμενη αξία. Και κοιτώντας τις επιπτώσεις των μέτρων που έχουν να κάνουν με την αναδιάρθρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα δούμε ότι υπάρχουν δύο όψεις σε αυτό το ζήτημα. Πρώτα, μία περίοδο από το, από το 1975 έως το 2002, όπου η Ευρωπαϊκή Ονομοθεσία δεν ασχολείται άμεσα με τα ζητήματα αναδιάρθρωσης, αλλά πολύ έμεσα για παράδειγμα την οδηγία για την πληροφόρηση και την συμβουλευτική, όπου γίνεται μια πολύ μικρή παραπομπή στην αναδιάρθρωση. Στο σημείο 9. Έπειτα, από το 2002 μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει νομική πρωτοβουλία πλέον. Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση μέσω της οποίας ε, διαπιστώνουμε ότι χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες πρακτικές ως κίνητρο για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης στις κοινωνικές επιπτώσεις και στις επιπτώσεις των χώρων εργασίας. Οι επιπτώσεις αυτών των δύο περιόδων στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες είναι ότι πράγματι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή δράση στον τομέα αυτό, αλλά υπάρχουν και δυσκολίες εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας στην ε, τωρινή κατάσταση. Η ισχύουσα οδηγία λοιπόν θα ήταν καλό να αναθεωρηθεί Υπάρχουν πολλές δυσκολίες στη δημιουργία ορισμού της αναρδιάρθρωσης και στην ε, προσμονή των αλλαγών. Επίσης υπάρχει κάποια ασάφεια ανάμεσα στις οδηγίες, για παράδειγμα την οδηγία για τις ε, συλλογικές συμβάσεις. Για παράδειγμα, από τους ε, τους αναδόχους. Μετά την περίοδο αυτή, 2002-2012, έχουμε δει ότι, έχει... ότι έχουμε λίγη έως ε, καθόλου πρόοδος. Και πιστεύουμε ότι αυτό επηρεάζει αρνητικά τους απασχολούμενους τους εργαζόμενους, καθώς και αρνητικά και τη δυναμική στις ε, περιφέρειες. Διότι η αναρδιάρθρωση μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένες περιφέρειες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα ήταν αυτά. Σε εθνικό επίπεδο, ας δούμε τι ευρήματα έχουμε. Υπάρχει μία όχι τόσο καλή εφαρμογή της, ε, κοινωνικής, της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Οδηγίας η οποία εν μέρει ασχολείται με την αναδιάρθρωση και την συμβουλευτική και την πληροφόρηση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί, όντως. Βέβαια, η αντιμετώπιση σε εθνικό επίπεδο της ε, κοινωνικής άποψης της ε, διεθνικής αναδιάρθρωσης είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και Επίσης εδώ παρατηρούνται ασυμμετρίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης παρατηρείται έλλειψη λογοδοσίας στο επίπεδο της επικουρικότητας. Εδώ παρατηρούμε ορισμένες δυσκολίες στην εφαρμογή της ε, οδηγίας για την εργασία καθώς φαίνεται το ζήτημα της ε, ευθύνης υπόκειται σε εθνικές οντότητες. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με το δίκαιο του ανταγωνισμού και εξετάζοντάς το θα δούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σύνδεσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σύνδεσης της οδηγίας με την λογοδοσία σε εθνικό και μη επίπεδο και σε επίπεδο αναδόχων. Εδώ στο τέλος της διαφάνειας θα δείτε έναν κατάλογο από ενδιαφέροντα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που χρηματοδοτούνται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ασχολούνται κυρίως με την αναδιάρθρωση, τα περισσότερα, με την ε, συμβουλευτική και την πληροφόρηση και την αντίστοιχη οδηγία. Εμείς αυτό που παρατηρούμε είναι τρία σημεία τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε εάν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση που ισχύει τώρα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στον τομέα της αναδιάρθρωσης όσον αφορά την πρόβλεψη των αλλαγών και την διαχείριση της αναδιάρθρωσης. Ο χρόνος και η εμπιστοσύνη. Ο χρόνος και η εμπιστοσύνη χωρίζονται σε, διαχεί ποιοτική διαχείριση του χρόνου, στην πρόβλεψη της αλλαγής. Εάν δηλαδή θέλουμε να προβλέψουμε και να προλάβουμε δραματικές ε, επιπτώσεις στον χώρο εργασίας, πρέπει να προβλέψουμε, πρέπει να κάνουμε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και αυτό να γίνει μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέλη, δηλαδή τους εργαζόμενους. Ε, γι' αυτό έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα όργανα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή τη συμβουλευτική και την πληροφόρηση και την αντίστοιχη οδηγία 2014. Θα δείτε ότι αυτά είναι σημεία κλειδιά στις διαπραγματεύσεις προς μια συλλογική συμφωνία και όχι μια μονομερή απόφαση. Κάτι το οποίο υπάρχει εν μέρη στην ισχύουσα οδηγία, αλλά κανείς δεν το παίρνει στο σοβαρά. Ένα από τα κύρια αποτελέσματα των project αυτών που άρχισαν το 2006 και τρέχουν μέχρι και τώρα είναι οι αρχές σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμερε και αναμειγμένε στην διαδικασία αναδιάρθρωσης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η... να ελεγχιστοποιηθούν οι δραματικές ε, επιπτώσεις που θα επιφέρει η αναδιάρθρωση. Έπειτα, η διεθνικότητα είναι ένα άλλο επίπεδο της ε, λήψης αποφάσεων και της διάδοσης πληροφοριών. Και τώρα περνάμε στην τελευταία διαφάνεια, την βελτίωση φυσικά. Η βελτίωση μπορεί να γίνει μέσω της ενίσχυσης των υπαρχόντων νομικών οργάνων, αλλά όχι μόνο και ο νομικός ακτιβισμός, ιδιαίτερα στα πλαίσια των ε, διεθνικών ε, συλλογικών συμβάσεων. Με τη μορφή προτάσεων και εδώ σε αυτή τη διαφάνεια μπορείτε να δείτε τα υπέρ και τα κατά, τις καλές και τις άσχημες πλευρές. Τα υπέρ είναι η μετάβαση από διμερή σε πολυμερή ανάμιξη και ανάληψη ευθυνών, κάτι που λείπει προς το παρόν. Η υπεύθυνη εταιρική διαχείριση, η πρόβλεψη της αλλαγής και η καινοτομία, η φροντίδα για την υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, η λογοδοσία και οι κυρώσεις, το δικαίωμα στην κατάρτιση και κάτι που λείπει και ελπίζουμε να δούμε στο μέλλον ε, ως, ε, με τη μορφή πρότασης είναι η αναδιάρθρωση στον δημόσιο τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο καθηγητής Άλλες από το Πανεπιστήμιο του Κασίνου στην Ιταλία έχει το λόγο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα μπορώ να μιλήσω εδώ στο βωμό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και θα εστιάσω στις νομικές πτυχές αυτής της ε, προοπτικής, της ε, νομοθετικής πρότασης. Το σχέδιο υπευλήθη τον Ιούνιο και βεβαίως υπάρχει πίεση χρόνου, οπότε θα απαντήσω στην ερώτηση που έχει τεθεί όσον αφορά αυτήν την ε, αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα είναι ε, αν μπορούμε καταρχήν να δούμε μια αντίθεση μεταξύ της νομοθετικής δράσης ή μη και δεύτερον μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου ή η υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μία από τις σημαντικές ε, ερωτήσεις που απορρέουν από αυτήν την ερώτηση είναι το ποια θα είναι η επιλογή παραδείγματο χάρη για μια οδηγία. Κατά την άποψή μου θα είχε συνοχή όσον αφορά την νομική βάση που έχει υιοθετηθεί σε αυτή την πρόταση να επιλεγεί η οδηγία. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει δεσμευτικός χαρακτήρας μία μη δεσμευτική, μη ρυθμιστική δραστηριότητα, όπως παραδείγματο χάρη ένας κώδικας διοντολογίας, θα μπορούσε να προστατεύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων, που αυτός είναι ο κύριος σκοπός αυτής της πρότασης τελικά. Δεύτερη υποερώτηση. Υπάρχουν ε, κάποιες άλλες ε, δυνατότητες ρυθμιστική δράση ή μη ρυθμιστική δράση. Κατά την άποψή μου, ένα μη δεσμευτικό νομικό πλαίσιο θα έχει αποτελέσματα μόνο και εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι στο επίπεδό τους έχουν υιοθετήσει ένα αυτορυθμιστικό εργαλείο. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να διαπραγματευθούν υπό τη σκιά και στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας και εάν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε μόνο ισχύει η οδηγία. Η προτινόμενη δράση μπορεί να ξεπεράσει αυτούς τους στόχους, εάν αυτοί θεωρούνται ικανοποιητικοί. Κατά την άποψή μου δεν είναι ικανοποιητική με την έννοια ότι εδώ ε, καθορίζουμε ένα ελάχιστο κοινά αποδεκτό πρότυπο και όπως έδειξε ο συνάδελφος, υπάρχουν πολύ διαφορετικές ρυθμίσεις από τη μία χώρα στην άλλη και υπάρχουν τελείως διαφορετικές πηγές. Συλλογικές συμβάσεις, διοικητικές ε, πηγές, νομοθετικές πηγές, είτε άλλου είδους ε, νομοθετικές πηγές. Τελικά λοιπόν βλέπουμε ότι η συνοχή αυτής της πρότασης και η επίτευξη του στόχου καθώς και η υλοποίηση είναι αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αν κοιτάξει κανείς τη δεύτερη σύσταση, διαπιστώνει ότι ο κύριος στόχος αυτής της πρότασης είναι η βελτίωση της ε, προετοιμασίας και της διαχείρισης με έναν ε, κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο μίας αναδιάρθρωσης με τη συμμετοχή των εταιριών, των εκπροσώπων των εργαζομένων, των κοινωνικών εταίρων. Και βλέπουμε ότι η οδηγία αυτή δεν έχει νομική βάση όσον αφορά αυτό τον κύριο στόχο. Και την ίδια ώρα είναι πολύ δύσκολο βάσει του άρθρου 153 ένα, να διαπιστώσει ότι υπάρχει κοινοτική αρμοδιότητα όσον αφορά την προετοιμασία, την πρόβλεψη και την διαχείριση μιας αναδιάρθρωσης. Προσπάθησα λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα, να εντοπίσω την, την προσοχή μου σε κάποιες εναλλακτικές στο άρθρο 153 ή σε κάποια άλλα σημεία της συνθήκης. Βεβαίως, είμαι στην Επιτροπή Απασχόλησης και η πρώτη επιλογή θα ήταν η καλύτερη. Το αρθρο 153 1 153.1β αναφέρει μία πολύ ευρή αρμοδιότητα στις συνθήκες εργασίας και στα πλαίσια αυτή τη αρμοδιότητα μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι εμπίπτει ο στόχος ε, της ε, οδηγίας αυτής. Βεβαίω υπάρχει και η δυνατότητα να αναφερθεί κανείς στο άρθρο 153.1.F όπου αναφέρεται και η συν απόφαση χωρίς όμως να αναφέρεται πουθενά ότι υπάρχει εδώ αρμοδιότητα κοινοτική και εδώ μπορεί κανείς να αναφερθεί στο άρθρο 352 όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων. Προφανώς υπάρχει εδώ βεβαίως και περιθώριο για εθνικές αποφάσεις. Και μπορείτε στην έκθεσή μου να βρείτε κάποια στοιχεία που αναφέρουν αυτές τις δυνατότητες. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε επίσης ότι εδώ δεν υπάρχει απολύτως καμία αναφορά στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές Εργαζομένων. Κατά την άποψή μου, ο στόχος αυτής της πρότασης δεν μπορεί να επιτευχθεί και σε καμία περίπτωση αυτές οι υποχρεώσεις οι οποίες επεριέχονται στην ομοθεσία κάποιων κρατών μελών καθώς και κάποια νομικά μέτρα τα οποία προβλέπονται για την περίπτωση αναδιαρθρώσεων. Τέλος και πολύ σημαντικό πέρα από αυτές τις επιπλέον υποχρεώσεις, αυτή η πρόταση δεν εμπεριέχει καμία προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις υπάρχουσες νομοθεσίες όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις. Και τώρα θα περάσω στη δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων, αυτών που έχουν σχέση με την συνοχή αυτής της πρότασης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Υπάρχει συνοχή με τα άλλα μέτρα, με τις άλλες πολιτικές Κατά την άποψή μου, όσα έχει η πρόταση αυτή, δεν είναι συνεκτική με τις άλλες ε, πολιτικές στον αντίστοιχο τομέα. Αν κοιτάξουμε το προήμιο, βλέπουμε ότι στην πρόταση αυτή δεν υπάρχει καμία αναφορά σε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός, κυρίως με κάποιες σημαντικά μέτρα και πολιτικές, όπως για την υγιεινή και την ασφάλεια, για τις συλλογικέ απολύσεις, διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις. Επιπλέον, η οδηγία αυτή θα πρέπει να περιέχει και κάποια σημεία συντονισμού με άλλα ε, κείμενα τα οποία μπορείτε να βρείτε, τα αναφέρω στην έκθεσή μου. Γι' αυτό και η απάντηση σε αυτή την ερώτηση σαφώς και εξαρτάται από την ε, τροποποίηση αυτής της πρότασης και από, την, από τον συντονισμό με την ήδη υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία αν υπάρξει συντονισμός, ναι, θα βελτιωθούν οι σύνθεκες εργασίας των εργαζομένων. Εάν υπάρξει συντονισμός, η πρόταση αυτή θα βελτιώσει το δικαίωμα σε ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων. Υπό αυτόν τον όρο, λοιπόν, ναι. Και κάτι άλλο που θεωρώ πολύ σημαντικό, μια άλλη ερώτηση, είναι σε ποιο βαθμό η πρόταση αυτή στηρίζει την προσέγγιση για περισσότερη ευελιξία και ασφάλεια. Πρόκειται για τις δυνατότητες που δίνονται σε επιχειρήσεις αλλά και σε εργαζόμενους να προσαρμοστούν καλύτερα στα δεδομένα ενώ αυξάνεται η εγγύηση και η ασφάλεια που δίνεται στους εργαζομένους. Συμπερασματικά θα ήθελα να πω ότι η πρόταση αυτή, ως έχει σήμερα, έχει κάποια ενδιαφέροντα δυνατά σημεία, κάποιες αδυναμίες και σαφώς χρειάζεται περισσότερο συντονισμός με την υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και ισχύοντα μέτρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Και τώρα να περάσουμε στο τέταρτο προσκεκλημένο μας, που είναι ο κύριος Ούσμαν Καν, που από το Ηνωμένο Βασίλειο και από το Matrix Insight. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση να έρθω και να σας μιλήσω σε αυτό το, αυτό το απόγευμα. Ήδη ακούσατε την ε, λογική που έχει να κάνει με αυτή την ε, προτινόμενη οδηγία και την νομική λογική της προτινόμενης οδηγίας, ενώ εγώ Τώρα θα σας μιλήσω για το εξής, να δούμε το οικονομικό, την οικονομική λογική που υποστηρίζει αυτή την προτινόμενη οδηγία και συγκεκριμένα να δούμε ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος της προτινόμενης οδηγίας. Σε ό,τι αφορά τη δουλειά που κάνουμε για τα ευρωπαϊκά όργανα και πέραν αυτών, θα ήταν ε, σχετικά απλή η ερώτηση, θα φαινόταν σχετικά απλό το ζήτημα, όμως μπορώ να σας πω ότι η ερώτηση είναι πιο απλή από την απάντηση. Και νομίζω ότι για μια στιγμή αξίζει να σκεφτούμε το γιατί. Γιατί θεωρήσαμε ότι είναι τόσο δύσκολο να δοθεί απάντηση σε αυτή την ερώτηση και υπάρχουν ε, δύο κυρία στοιχεία εδώ τα οποία σχετίζονται με τα δεδομένα και την έρευνα. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα δεδομένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την ανεργία και με την απασχόληση. Αλλά η διαθεσιμότητα των δεδομένων σε σχέση με την προτινόμενη αναδιάρθρωση και την πραγματική αναδιάρθρωση και την προτινόμενη κατάρτιση και την πραγματική κατάρτιση ουσιαστικά είναι πολύ λιγότερο από ό,τι για άλλους τομείς και θα αναφέρουμε στη συνέχεια ποιο είναι το σημείο αφετηρίας ε, και έχει γίνει προσπάθειες να υπάρξει μια βάση εργασίας, όμως μπορεί να υπάρξει και μια δυνατότητα απασχόλησης. Επίσης, σε σχέση με την αξιολόγηση του αντικτύπου. Θα θέλαμε να έχουμε ε, ερευνητικές μελέτες που θα εξετάζουν τις συνέπειες ε, της έγκαιρης διαβούλευσης και κατάρτισης. Υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες και μπορούσαμε να τις λάβουμε υπόψη. Όμως και πάλι, αν δείτε άλλους τομείς ε, για την απασχόληση και ε, ευρύτερους τομείς κοινωνικής πολιτικής, πρέπει να πούμε ότι η ποιότητα και το εύρος των μελετών ε, δεν είναι τόσο καλό όσο θα περίμεναν κάποιοι. Και επίσης, ε, αν σκεφτούμε το τα πιθανά ωφέλη ε, θα ήταν ε, να αποφύγουμε τις απολύσει ή να ε, ξαναφέρουμε τους εργαζομένους σε θέσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν μιλάμε για μεδέτικη 20.000 ευρώ ετησίως ε, που καταβάλλονται σε επίδομα ανεργίας. Ε, έτσι λοιπόν, αν κάποιος μπορεί να ξαναβρει δουλειά τρεις μήνες νωρίτερα, ε, αυτό θα ήταν καλό. Και έτσι λοιπόν, σε σχέση με το πιθανό όφελος, υπάρχει σημαντικό όφελος, αλλά σε σχέση με την βάση των επιδεκτικών στοιχείων θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί. Τι κάναμε εμείς, μπορέσαμε να βρούμε και δεδομένα και μελέτες έρευνας, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να γίνει μια απλή σύνδεση μεταξύ της έγκαιρης διαβούλευσης και της κατάρτισης και της ε, ασφάλειας ε, στην εργασία και της απασχολησιμότητας. Εδώ Βλέπετε σε αυτό το διάγραμμα ότι κυρίως εξετάσαμε τις συνέπειες της έγκαιρης διαβούλευσης για την απασχολησιμότητα και την ε, συνέπεια της κατάρτισης στην ασφάλεια ε, της διατήρησης της εργασίας και προσπαθήσαμε να δούμε αν υπάρχει διασταυρούμενη επιρροή στα στοιχεία αυτά. Λοιπόν, οι λεπτομέρειες είναι στην έκθεση, αλλά για να συνοψίσω, τα συμπεράσματα της μελέτης, εμείς ε, μπορέσαμε να πούμε ότι αν δείτε τις διαθέσιμες μελέτες ε, και τα δεδομένα που υπήρχαν εκ των προτέρων, διεφάνει ότι όπου υπήρχε έγκαιρη διαβούλευση και κατάρτιση, ήταν θετικό ο αντίκτυπος και στην ασφάλεια διατηρήσης της ενεργασίας και στην απασχολησιμότητα. Πρέπει να πω εδώ κάτι σημαντικό, ότι εμείς μπορέσαμε να δούμε τον πριν και το μετά. Ε, αυτό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να δούμε ποιες είναι οι αιτίες, ποιες είναι η αιτιότητα. Να πούμε, η έγκαιρη διαβούλευση και η κατάρτιση προκάλεσαν αυτό τον αντίκτυπο. Όμως ε, κάνουμε την ε, υπόθεση ότι υπήρξε ο αντίκτυπος αυτός. Τώρα, θα αναφερθώ σε δύο τομείς. Ε, καταρχήν, ε, να δούμε τι συμβαίνει σε επίπεδο επιχείρησης ε, και σε λίγο θα δούμε τον πανευρωπαϊκό αντίκτυπο. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε σε αυτό το πρώτο διάγραμμα. Να μπορούμε να πούμε ότι βάσει των μελετών που εξετάσαμε και, τα δεδομένα, και βάσει των δεδομένων που είχαμε, θέλαμε να μπορέσουμε να πούμε το εξή ότι αν εισαγόταν αυτή η οδηγία, σε ποιο επίπεδο θα έπρεπε να έχει αντίκτυπο στην απασχόληση για να έχουμε μια καλή σχέση κόστους-οφέλους και στα περιθώρια. Λέμε ότι αν μπορεί κανείς ε, να εξοικονομήσει το 60% των ε, αρχικά προτινόμενων απολύσεων μέσω της έγκαιρης διαβούλευσης, τότε θα λέγαμε ότι έχουμε καλή σχέση κόστους αποτελέσματος. Τώρα, αν δείτε το αποτέλεσμα της μελέτης, ε, λέμε ότι τα νούμερα ήταν πάνω από αυτό το επίπεδο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει εσείς να επικεντρωθείτε σε αυτά τα υψηλά αριθμητικά στοιχεία, αλλά πρέπει να δείτε το σημείο της αλλαγής, για να μπορεί να πει κανείς σε ποιο σημείο θα ωφελούσε το κόστος και πού έδειξε η μελέτη ότι επιτέχθη ε, αυτή η εξοικονόμηση του κόστους. Τώρα, αν δούμε τι συμβαίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο στη μελέτη μας. Όπως ε, θα γνωρίζετε, σε εθνικό επίπεδο, σε ορισμένα κράτη-μέλη, ήδη υπάρχει εθνική νομοθεσία που καλύπτει τις διατάξεις ε, που καλύπτει αυτή η προτινόμενη οδηγία. Έτσι λοιπόν θα αναμένατε ότι ο αντίκτυπος της οδηγίας ε, σε επίπεδο εταιρείας ε, θα ήταν ουσιαστικά πρέπει με πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ βλέπετε έχουμε μια, ένα κατάλογο χωρών από το α στο σιγματάφ A μέχρι F. Εδώ θέλαμε να δούμε τα σημερινά επίπεδα και της διαβούλευσης αλλά και της κατάρτισης και να βασιστούμε σε αποδεκτικά στοιχεία για να μπορέσουμε να ταξινομήσουμε τα κράτη-μέλη που ε, παρουσιάζουν ε, επιδόσεις υψηλές, ε, μέτριες ή χαμηλές. Και κατόπιν θέλουμε να δούμε ποιος θα ήταν ο συνολικός αντίκτυπος στα 27 κράτη-μέλη. Και το πόρισμα είναι ότι ο συνολικός αντίκτυπος θα ήταν στο επίπεδο περίπου του 50% του αντίκτυπου που θα βλέπαμε σε μία συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό λοιπόν για να πούμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη ήδη υπήρχαν διατάξεις ε, που κάλυπταν ε, την οδηγία σε σχέση με τη διαβούλευση και την κατάρτιση. Αυτό που μας ζητήθηκε να κάνουμε και μας ε, ζητήθηκαν αυτέ οι μελέτε για να καλύψουμε διάφορες περιπτώσεις και διάφορες οργανώσεις. Όμως για πρώτη φορά προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε αυτά τα διάφορα μέρη ως προς την εξέταση του αντικτύπου. Και υπάρχει ένα σημαντικό πεδίο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια μελλοντική δουλειά. Δηλαδή όχι μόνο να ενδυναμώσουμε ε, τη βάση των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά θέλουμε να βελτιώσουμε και την ποιότητα και την ποσότητα και την αξιοπιστία της συλλογής των δεδομένων. Θεωρούμε ότι αυτός θα είναι ένας εξαιρετικός στόχος, δηλαδή να ενδυναμώσουμε τη βάση των δεδομένων και να προωθήσουμε και την βάση την ερευνητική. Εδώ υπάρχουν κάποιες πτυχέ που θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να βελτιωθούν πέραν αυτών. Θεωρούμε ότι η μεθοδολογία που θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε είναι ένα σημαντικό σημείο αφετηρίας. Και τουλάχιστον στο επίπεδο αυτό μας δίνει μία ένδειξη ότι θα μπορούσε να υπάρξει σημαντικός θετικός αντίκτυπος ε, της προτινόμενης οδηγίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτές οι τέσσερις παρουσιάσεις δείχνουν ότι για ένα τέτοιο σημαντικό θέμα όπως αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της έκθεσης πρωτοβουλίας, μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να ακούμε εμπειρογνώμονες, να ακούμε ειδικού, οι οποίοι γνωρίζουν την κατάσταση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και το πώς μπορεί κανείς να προοδεύσει κάτι που σίγουρα θα το λάβει υπόψη του ο εισηγητής. Ξεκινάει η συζήτηση. Ο εισηγητής έχει το λόγο και και ο εισηγητής. Δηλαδή έχω 10 λεπτά αυτό μου λέτε. 30 δευτερόλεπτα θα μίλησω. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τους τέσσερις ομιλητές. Δεν ε, είχα χρόνο να διαβάσω το σύνολο της τεκμηρίωσης, αλλά πρέπει να είστε βέβαιοι καταρχήν ε, για το ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο έργο μας. Και εγώ πιστεύω ότι πέρα από το έργο αυτής της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας, νομίζω ότι μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι εδώ αυτό θα αποτελέσει ένα λίθος στην οικοδόμηση μιας καλύτερης Ευρώπης. Ε, πρόκειται για ένα εγχείρημα ε, το οποίο είναι αξιοσημείωτο και από νομική σκοπιά, από οικονομική, από κοινωνική σκοπιά και όπως είπατε και εσείς απευθυνθήκατε στον οίκο που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες και μας είπατε πώς έχει κατάσταση, ποιο είναι το πρόβλημα και ποιες θα μπορούσε να είναι η λύση. Είναι, απαιτητική, είναι απαιτητικό αυτό το εγχείρημα και μάλιστα είναι πολύ πιο απαιτητικό ε, στους ε, ακαδημαϊκές ε, στα ακαδημαϊκά πλαίσια, όμως είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στα καθήκοντά μας τα οποία θα πρέπει να τα αναλάβουμε θέλοντας και εμεί. Γιατί αυτό το θέμα των αναδιαρθρώσεων ουσιαστικά το βλέπουν πολύ λανθασμένη προοπτική. Θεωρούν ότι ε, υπάρχουν ε, θέματα ιδεολογικά, αιτιολογικά, όχι. Κοιτάξτε, ε, αυτό το θέμα γίνεται επιτακτική ανάγκη και είτε θα το κάνουμε καλύτερα στο μέλλον ή θα συνεχίσουμε ε, όπως δρούμε σήμερα. Και αν το κάνουμε αυτό, η Ευρώπη θα βρεθεί σε μια καταστροφή, θα έχει καταστρέψει τα βιομηχανικά της δίκτυα και θα έχει ε, καταστραφεί η διάρθρωση της κοινωνίας μας ε, και βλέπουμε με τι ταχύτητα κινούνται αυτές οι διαδικασίες, βλέπουμε μέσα σε 100 χρόνια πώς καταστρέφονται οι αξίες που έχουμε συσσωρεύσει στην Ευρώπη. Είδαμε την ε, συνέβη και με την ε, Arsenal Metal ε, και χάνουμε γνώση, καταστρέφεται μια ολόκληρη κοινωνία. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω αν σήμερα θα καταρθώσω να πείσω τους συναδέλφους ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να νομοθετήσουμε και να αναλάβουμε δράση. Σίγουρα, πάντως, ε, όλα αυτά που ακούστηκαν δεν θα είναι άχρηστα. Μας ε, βοηθήσατε πάρα πολύ να καταλάβουμε για να προωθήσουμε την αλλαγή αν ε, μου επιτρέπετε, ε, έλεγε ο Καρλός Μάρξ ότι το καθήκον μας είναι να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να τον γνωρίσουμε τον κόσμο για να τον αλλάξουμε και φυσικά η δική σας δουλειά μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τον κόσμο και ε, εγώ είμαι ικανοποιημένος και για τις κριτικές και για τους επένους που ακούστηκαν για την εκθεσή μου, γιατί θα μας βοηθήσει στην αλλαγή. Πραγματικά αισθάνομαι ανακούφιση γιατί νομίζω ότι και εγώ και οι συνάδελφοί μου κάνουμε ένα λογικό εγχειρήμα και προσπαθούμε εδώ να πράξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να μην ακρηγορήσω, θα ήθελα να κάνω μια γενική ερώτηση σε όλους σας και μια συγκεκριμένη ερώτηση που με ανησυχεί πάρα πολύ και κυρίως θέλω να απευθυνθώ στον καθηγητή Εντοάρντο Άλες και νομίζω ότι έθεσε όχι μόνο πολιτικά αλλά και τεχνικά και νομικά προβλήματα και θα του κάνω κάποιες ερωτήσεις γιατί πρέπει να βελτιώσει την εκθεσή μου προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρώτη ερώτηση γενικού χαρακτήρα. Αναφερθήκατε στη συνοχή που θα έπρεπε να έχει αυτό το νομοθέτημα με το σύνολο ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών. Μιλήσατε για την ευελιξία και ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να επανέλθουμε εκεί, γιατί έχουμε μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα όπου έχουμε κάθε ευελιξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά δεν δίνει καμία ασφάλεια γιατί υπάρχουν κάποια παθητικά υποκείμενα αυτών των ευέλικτων πολιτικών και αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ με την οδηγία μου είναι να δώσω νόημα σε αυτά τα λόγια της ευελιξίας και ασφάλειας. Δηλαδή να μην έχουμε μόνο ευελιξία αλλά και ασφάλεια. Αλλά δεν μιλώ για τη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Θα θέλαμε να μου πείτε η συνοχή που υπάρχει με τους μεγάλους στόχους ε, που τίθενται στα έγγραφα της Ένωσης, στις αποφάσεις του Συμβουλίου και της ε, Κομισιόν. Ε, μιλάνε για αριστεία. Είναι ε, ουσιαστικά συνεκτικό αυτό το έργο. Δηλαδή δίνεται να έχουμε πιο αποτελεσματικά οικονομικά αποτελέσματα και θα φτάσουμε στην Ευρώπη του 2020 και να αφήσουμε το Λεσέφερ που αφήνουμε σήμερα. Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι και για τους τέσσερις. Να μου πείτε, για μένα, θέλω να μου πείτε αν υπάρχει συνοχή, γιατί για μένα είναι πολιτικά σημαντικό αυτό. Είδαμε τι αναφέρεται στην ανακοίνωση τη Κομισιόν, αλλά αυτά έχουν σχέση ή δεν έχουν σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική. Η συγκεκριμένη ερώτηση που με απασχολεί είναι ότι υπάρχουν κάποια συνάδελφοι που δεν βλέπουν κάτι που για μένα είναι προφανέ. Θέλω να μου εξηγήσετε και να μα πείτε Ποια αξία δίνετε εσείς στο να καθερώσουμε το δικαίωμα για την κατάρτιση, ότι ε, πρέπει οι εργαζόμενοι να καταρτήσονται με τον κατάλληλο τρόπο για την πρόβληψη και τη διαχείριση των τεχνολογικών αναγκών. Εγώ ε, θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ένα δικαίωμα που δίνεται εις βάρος ε, της ε, ικανότητας των επιχειρήσεων. Το αντίθετο μάλιστα είναι για να γίνουν πιο ικανές επιχειρήσεις μας για να κερδίσουν το μέλλον. Και τέλος, στρέφομαι κυρίως ε, στον κύριο Άλες, τον Ιταλό καθηγητή, γιατί ε, υπάρχουν κάποια ισχυρά και κάποια δύναμα σημεία, αλλά θέλω να μου απαντήσετε, γιατί είναι αλήθεια ότι μια μικρή έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας, εγώ δεν μπόρεσα να επιλύσω όλα τα προβλήματα που μπορεί να θέτει η συνοχή αυτού του νομοθετήματο με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά πρέπει να σας πω κύριε καθηγητά, αλλά δεν ε, είναι οδηγία αυτή ακόμη. Γι' αυτό η ερώτησή μου είναι, εσείς πιστεύετε αυτά προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή να βρούμε ε, την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αυτή τη οδηγία και των άλλων ε, νομοθετημάτων και είναι το κοινοτικό κεκτημένο σε μια μετέπειτα στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Αξίζει να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, ακόμη και αν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε, συνοχή και συμβατότητα τη οδηγίες αυτή με τι προηγούμενε. Ή πιστεύετε ότι είναι ένα δύνατο εγχείρημα από νομική σκοπιά. Και καθώς ε, έκανα αυτήν την ερώτηση, να πω και κάτι ακόμη. Εσείς ε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί στην πρόταση και τι δεν θα έπρεπε να αφήσουμε στη μέση σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, τι μπορώ να αφήσω στις μου και στη λογική που υπάρχει σε αυτό το Νίκο. Γιατί θα έπρεπε να θυσιάσω κάποιες από τις θέσεις μου. Και τι δεν θα έπρεπε να θυσιάσω υπό τον κίνδυνο να αποδυναμωθεί η πραγματική φύση και αυτή η θετική πτυχή που εσείς μας παρουσιάσετε εδώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λόπε Φαντανιέ. Σας ευχαριστώ όλους. Καταρχήν θα είμαι πιο σύντομη από το συνάδελφο. Θα ήθελα καταρχήν να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω γιατί νομίζω ότι το έργο σας είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα τόσο σημαντικό που πιστεύω ότι θα πρέπει να το μελετήσουμε εις βάθος. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι σε θέση να σας θέσω συγκεκριμένες ερωτήσεις, ε, πέρα από αυτές ε, που έκανα ήδη ο συνάδελφος, ο κ. Σέρκας. Γιατί εγώ νομίζω ότι το πρώτο που θα πρέπει να γίνει είναι να μελετηθεί εις βάθος η μελέτη που μας παραδώσατε. Νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε, δεν θα έλεγα ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τον κόσμο, ούτε θα μιλούσα για τον Μάρξ, γιατί πολλοί δεν ε, σκεφτόμαστε με τους όρους αυτούς, όμως εγώ νομίζω ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τις επιχειρήσεις, και τη σημερινή οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων αλλά και τι συνθήκε για του εργαζόμενου. Και είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να μπορούμε να εργαζόμαστε. Θα μα κοστίσει αυτό. Εγώ δεν ξέρω πώ θα φτάσουμε στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου, γιατί βλέπω όλο ένα να γίνεται πιο πολύπλοκη η κατάσταση και ότι πρέπει να διαπραγματευόμαστε όλο ένα και περισσότερο και θέλουμε να έχουμε ένα κείμενο καλό για όλου που να χρησιμεύει για όλε τι χώρε. Γιατί κάτι που δεν είναι για μένα σαφές, για το οποίο έχω αμφιβολίες αν θέλετε, είτε μιλάμε για οδηγία είτε για σύσταση. Εγώ νομίζω ότι ε, τα κράτη-μέλη δυστυχώς αν δεν θέλουν να εφαρμόσουν μια οδηγία δεν θα το κάνουν. Το θέμα είναι πώς θα τις εφαρμόσουν τις βελτιστές πρακτικές και πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και να μελετηθεί σε όλες τις χώρες τι εφαρμόζεται και μη. Εγώ νομίζω ότι και αναφέρθηκε από όλους τους ομιλητές ότι υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των διάφορων χωρών και δεν είναι σαφές για μένα το πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τουλάχιστον κάποιες ελάχιστες βελτιστές πρακτικές προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Και να επαναλάβω ότι θα σας καλέσω για να σας θέσω συγκεκριμένες ερωτήσεις αφού θα μελετήσω λεπτομέρως τα έγγραφα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ποιο άλλο ήθελε να πάρει το λόγο. Ο κύριο Χέντελ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση για τους εμπειρογνώμονες, διότι δεν άκουσα τίποτα πάνω σε αυτό. Και θα ήθελα να το αναφέρω, διότι πιστεύω το παράδειγμα των βέλτιστων πρακτικών δεν αναφέρθηκε εκτενώς από τους εμπειρογνώμονες. Εμείς στη Γερμανία έχουμε μία ιδιαίτερα ανεπτυγμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης και αλλαγής στον επιχειρησιακό χώρο και ως προς τις μαζικές απολύσεις και την αποφυγή τους και αγγίζοντας άλλους τομείς και ε, ως προς την ενημέρωση και των εργαζομένων και των εργοδοτών. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι όσον αφορά την ε, αναδιάρθρωση η Γερμανία εξαιτία της αναδιάρθρωσης ε, αναμενόταν να υποφέρει στον εργασιακό χώρο, αλλά συνέβη το αντίθετο. Ως 25 χρόνια διετέλεσα επικεφαλής ενός συνδικάτου στη Γερμανία και ασχοληθήκαμε εκτενώς με την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, την ασφάλεια των εργαζομένων και ήμασταν αρκετά επιτυχείς στο έργο μας. Ε, επομένως δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε να κάνουμε λόγο για βάρος και κόπο που επιφορτίζεται ο εργοδότης, αλλά το αντίθετο μάλιστα. Στη Γερμανία οι εργαζόμενοι μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα απαντώνται οι απορίες τους και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να μπορούν οι εργαζόμενοι να είναι σίγουροι ότι θα έχουν επαρκή πληροφόρηση και αντιπροσώπευση. Ε, θα έλεγα θα πρότεινα μάλλον να καλέσουμε εδώ προσωπικά τους ε, αντιπροσώπους των εργοδοτών και εάν γίνει αυτό σας εγγυώμαι ότι θα βρεθούν τουζίνες από, από μάνατζερ οι οποίοι θα είναι θετικοί προς ε, την ε, διαδικασία αναδιάρθρωσης, προς, πως δεν θα αρνηθούν, διότι με αυτόν τον τρόπο και τα δικά τους συμφέροντα και η δική τους ε, ασφάλεια προς το μέλλον θα μπορέσει να διασφαλιστεί. Αυτό είναι παράδειγμα καλών πρακτικών για την Ευρώπη. Αυτό θα ε, προσέδιδε προς τη θεμενή αξία στην Ευρώπη. Όχι μόνο η ανάλυση δεδομένων, αλλά και η ανάμειξη των ε, παραγόντων, των ενδιαφερομένων στη διαδικασία. Εγώ ήμουν επί 25 χρόνια ενεργός στον τομέα αυτό και πιστεύω ότι και η ατομική και η συλλογική κατάρτιση είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τις ε, γερμανικές επιχειρήσεις διότι αυτό διασφαλίζει και την μετέπειτα εξέλιξη. Ανεργεί προς το συμφέρον και των δύο ε, μερών και αυτό στον τομέα της ε, αναδιάρθρωσης, εάν εφαρμοστεί, θα, είναι, θα έχει κέρδος και για τους δύο. Δεν θα τίθεται το θέμα ανταγωνισμού, αλλά θα βοηθούσε στην ε, περαιτέρω εξέλιξη. Πιστεύω πως αυτή η πρωτοβουλία είναι εξαιρετική του κυρίου Σέρκας. Αυτό που άκουσα από κάποιον αυτό που μπορώ να καταλάβω από αυτά που υπόθηκε, ναι, βέβαια είναι μια ε, έκθεση πρωτοβουλία, ναι, βέβαια πρέπει να ενωθεί και με άλλες ε, δράσεις και με άλλες πρωτοβουλίες. Πάντως αυτό που πρέπει να παραδεχτώ είναι ότι είναι ένα εξαιρετικό έργο, όμως η όλη διαδικασία δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο σε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, αλλά σε μια σύσταση ή ακόμα και σε μια οδηγία. Αυτό μπορούμε να αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό μπορούμε και πρέπει να κάνουμε εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης, να ασχοληθούμε ενεργά με αυτό το ζήτημα έτσι ώστε να ε, μπορέσουμε να θεσπίσουμε ολοκληρωμένους κανόνες και για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ποιος άλλος θα ήθελε το λόγο. Δεν βλέπω κανέναν. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους ομιλητές θέλει να αντιδράσει σε κάτι που άκουσε. Έχετε το λόγο. Βλέπω ότι θέλετε να μιλήσετε. Ευχαριστώ. Έχω πέντε λεπτά. Θα ήθελα να απαντήσω σε μία γενική ερώτηση του εισηγητή όσον αφορά την ύπαρξη συνοχής αυτής της πρωτοβουλίας με την ευελιξία και ασφάλεια, το flexicurity. Νομίζω ότι αν ακούσατε την παρουσίασή μου, είδατε ότι αυτή είναι μία από τις προστιθέμενες αξίες αυτής της πρότασης, με την έννοια ότι υπάρχουν υποχρεώσεις και για τους εργοδότες και για τις ε, δημόσιες αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να έχουν μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά το βαθμό ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Αλλιώς υπάρχει απλώς ευελιξία και όχι ασφάλεια. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε αυτήν την πτυχή ασφάλειας αυτής της διαδικασίας. Τώρα, το δικαίωμα για κατάρτιση, ναι. Αυτό όμως το θέμα είναι λίγο περίπλοκο με την έννοια ότι δεν πρέπει να το δούμε μόνο από την μορφή επιβολής ενός βάρους στις επιχειρήσεις. Πρέπει να το δούμε και σαν υποστήριξη αυτής της κατάρτισης μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ή της ε, δημόσιας παρέμβασης. Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά σημεία, τα δυνατά σημεία της πρότασης. Το θέμα τώρα του αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί ναι ή όχι. Να βελτιωθούν οι νομικές πτυχές. Δεν πρόκειται για οδηγία. Πρόκειται για πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Τώρα, νομίζω ότι αν διαβάσετε ε, τις σημειώσεις μου που υπάρχουν στο φάκελο που πρέπει να σας έχει μοιραστεί, λειτουργούμε βάση της αρχής ενημέρωση-διαβούλευση. Υπάρχει δηλαδή μια δυνατή βάση. Και πάνω σε αυτή τη βάση μπορούμε να θεμελιώσουμε τα επόμενα βήματα που ουσιαστικά έχουν άμεση σχέση με την συναπόφαση. Και εδώ έρχομαι σε αυτά που είπε ο Γερμανός ε, συνάδελφος, ε, Γερμανός βουλευτής. Ναι, μίλησα για βάρος, για υποχρέωση, με την έννοια ότι έτσι είχε τεθεί η ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι η γερμανική συναπόφαση με τη μία ή την άλλη προσέγγιση υπογραμμίζει ουσιαστικά αυτή την πρόταση. Κατά την άποψή μου, αυτό σίγουρα θα έδινε περισσότερα πλεονεκτήματα. Η αναδιάρθρωση σαφώς και μπορεί να υποφεληθεί από την συναπόφαση. Δεν είμαι κατά, είμαι 100% υπέρ και θεωρώ ότι οι επιδόσεις των ε, γερμανικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια είναι η απόδειξη ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Que... Θα ήθελε κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση για την κατάρτιση, δικαίωμα στην κατάρτιση. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σαφώς όλοι είμαστε υπέρ του δικαιώματος σε κατάρτιση. Δεν μπορεί κανείς να πάρει το λόγο και να πει ότι είναι κατά. Άκουσα τον συνάδελφο από την Matrix όσον αφορά την ασφάλεια των θέσεων απασχόλησης και θα ήθελα να πω για την κατάρτιση στην Ευρώπη, να σας δώσω κάποια στοιχεία. Όπως είπα και προηγουμένως, πώς αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις την αναδιάρθρωση, είναι κάτι που πολλές φορές δεν μας δείχνει στην πράξη τι κάνουν. Μία μελέτη που έγινε στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα το 2010 για τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη, στην ερώτηση έχετε κάποια κατάρτιση από τους εργοδότες σας, Σα έχει προσφερθεί κάποια κατάρτιση. Η απάντηση ήταν 37% ναι. Και σε πολλές χώρες τα ποσοστά ήταν πολύ χαμηλότερα. Αυτό πραγματικά μας δείχνει ποια είναι η πραγματικότητα όσον αφορά το δικαίωμα για κατάρτιση. Ναι. Έχετε το λόγο. Εν έχουμε την δυνατότητα τότε ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον αφορά για το δικαίωμα της ε, κατάρτισης και το καθήκον της ε, παροχής κατάρτισης. Πιστεύω πως εδώ το σημαντικό στοιχείο της πρότασης είναι η πρόσβαση στην ε, εκπαίδευση και στην κατάρτιση και η θεώρησή τους ως δικαίωμα. Είναι μια ευρωπαϊκή αξία και αυτή τη βασία έχει μέχρι τώρα. Δεν θα έπρεπε να θεωρείται καθήκον. Ιδιαίτερα αν δείτε την πρόταση θα δείτε ότι υπάρχει μία ε, κοινή πρόβλεψη για το ποιες θα είναι οι ανάγκες για κατάρτιση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και αν συσχετίσετε και αν συνδέσετε τους ε, ενδιαφερόμενους με αυτό, τότε το καθήκον της κατάρτισης θα γίνει καθολικό και όλοι θα είναι διαθέσιμοι να το παρέχουν και αυτό θα θέλαμε να το δούμε σε αυτήν την πρόταση. Τώρα όσον αφορά το αν χρειαζόμαστε ακτιβισμό νομικό στην αναδιάρθρωση. Πιστεύω ότι τα στοιχεία που έχουμε αποκομίσει από πολλές μελέτες δείχνουν ότι η αναδιάρθρωση γίνεται, εξελίσσεται σε ένα μόνιμο οικονομικό όργανο με πολύ σημαντικές επιπτώσεις, όπως ανέφερα στην αρχή, ε, για τους ε, εργαζόμενους, ε, για τους μισθούς, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για, το δημογραφικό ζήτημα. Εάν καταφέρουμε και, και αντιμετωπίσουμε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα με συνεκτικό και ολοκληρωμένο και λεπτομερή τρόπο, τότε πιστεύω ότι η μορφή μια οδηγία θα ήταν ο κατάλληλο τρόπο για να το πράξουμε, διότι μια οδηγία θέτει ελάχιστα πρότυπα. Και θα δώσει μια βάση για τα κράτη που δεν έχουν μέχρι τώρα νομική βάση σε αυτά τα ζητήματα. Έτσι λοιπόν ένα κράτος μέλος το οποίο έχει ε, ανώτερα πρότυπα όσον αφορά την ε, πληροφόρηση, διαβούλευση και την ε, πρόβλεψη ε, της αλλαγής δεν θα υποφεληθεί από μια οδηγία, όμως θα υποφεληθούν τα άλλα κράτη που δεν έχουν αυτά τα ελάχιστα πρότυπα ή που έχουν δυσκολία στην εφαρμογή των υπαρχόντων νομικών προτύπων. Το ίδιο επιχείρημα επανέρχεται ελάχιστη εναρμόνιση. Κύριε Κάν, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Όχι. Ωραία. Τελειώσαμε λοιπόν με το σημείο αυτό της συζήτησης. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί είναι η πρώτη φορά που και με αυτά τα πολύ σημαντικά επιχειρήματα μπορέσαμε να εξετάσουμε κάποιες πτυχές αυτού του θέματος. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε κάποιες από τις πτυχές της συζήτησης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Ο εισηγητής για το επόμενο σημείο. Είναι η παρουσίαση των τροπολογιών, των συμβιβαστικών τροπολογιών. 418 τροπολογίες έχουν υποβληθεί. Όπως είπατε μόλις, Πρόεδρε, υποβλήθησαν 419 ε, τροπολογίες Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο προκατακτικό στάδιο. Όπως βλέπετε από τον αριθμό των τροπολογιών και των αναλύοντε βάθο τροπολογίες, πράγματι υπάρχει μια πολυπλοκότητα, υπάρχουν και πολιτικά αλλά και τεχνικά προβλήματα. Εγώ ήδη προετοίμασα και με τους Σκιώδης ε, είχαμε μία πρώτη σειρά επαφών για αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες, είναι 16. Και νομίζω το 80% των ε, τροπολογιών έχουν ε, συμπεριληφθεί, καθώς είναι στοιχεία σχετικά ή στοιχεία που αφορούν την ευελιξία του κειμένου, να εμβαθύνουμε σε ορισμένα στοιχεία και πρόκειται για θέματα που δεν ε, θα θίξουν μια δεύτερη προσέγγιση. Δεν θίγουν δηλαδή τα πιο πολύπλοκα σημεία της συζήτησής μας. Εγώ νομίζω ότι η πρώτη απόφαση που λάβαμε ήταν ε, να πάρουμε περισσότερο χρόνο, καθώς ε, χρειάζεται να διαβάσουμε και να συζητήσουμε εις βάθος και επειδή υλοποιήσαμε και μόλις ε, αυτό το εγχείρημα, θέλαμε να ακούσουμε σχετικά με την προστέμενη αξία και τον αντίκτυπο που θα έχει η έκθεση αυτή καθ' αυτή και κάθε τμήμα της έκθεσης από νομική σκοπιά και πολιτική σκοπιά και στην πρώτη συνεδρίαση φτάσαμε μέχρι την σύσταση 6 αλλά θα πρέπει να κάνουμε όλο αυτό το εγχείρημα αφού θα έχουμε διαβάσει το σύνολο των στοιχείων που είναι επιτάπητος. Όπως και να έχει, για να ενημέρωσω τους συναδέλφους, εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξο ε, με τη δουλειά που έχει γίνει, γιατί προκύπτει ε, με σεφήνει ότι αν αφήσουμε κατά μέρου αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον ε, οίκο, αν αφήσουμε δηλαδή τις ευρωσκεψιστικές κατά μέρο, εγώ νομίζω ότι έχουμε σημαντική συνένεση μεταξύ μας ότι ήδη έχουν, έχει υπάρξει σημαντική καθυστέρηση. Ήδη έχουμε πολλά επιχειρήματα τα τελευταία 12 χρόνια που έχουν αναλυθεί και μελετηθεί για να, δώσουμε, για να κάνουμε ένα βήμα προς προστά και να υπάρξει ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία. Αυτό ήδη ήταν γνωστό γιατί επιλέξαμε ε, το 200... 28 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο εξή. Τι είδου νομοθετική πράξη θα μπορεί να ολοκληρωθεί με το εγχείρημα αυτό, θα είναι δεσμευτική πράξη ή μη δεσμευτική. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα, συνάδελφοι, και νομίζω ότι εμείς ε, θα πρέπει όλοι να κάνουμε ένα υπεύθυνο έργο, ανάλογα με το ότι είμαστε διατεθειμένοι να οικοδομήσουμε και μέχρι πόσο θέλουμε να προχωρήσουμε. Εγώ νομίζω ότι το σημερινό, η σημερινή συζήτηση και η συζήτηση που είχαμε και τις τελευταίες εβδομάδες θα μας βοηθήσει και εμπιστεύομαι στο ότι αυτό το κοινοβούλιο θα συνεργαστεί με τα εθνικά κοινοβούλια ε, και θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αντίληψή μας ε, για να δώσω ένα παράδειγμα για το τι ζητώ. Εγώ από την ε, δική μου έκθεση έχω αποσύρει το εξή. Έχει δύο τμήματα η έκθεσή μου και το πρώτο τμήμα θα ολοκληρωθεί στο τελευταία στιγμή της συζήτησή μας που θα αποφασίσουμε το στις πράξεις, αλλά στο δεύτερο τμήμα ε, είτε πρόκειται για δεσμευτική ή μη πράξη, όπως και να έχει πρέπει να μιλήσουμε για την αναδιάρθρωση. Εγώ νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μου, Πρόεδρε, και αυτό αφαίρεσε σε πολλές προβλήψεις, ε, να μπορέσουμε να συζητήσουμε ανεξάρτητα με το ποια οδό θα ακολουθήσουμε στο τέλος. Και εγώ στις συμβαστικές μου τροπολογίες, σε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες, έχω διαγράψει κάθε αναφορά για το αν θα είναι οδηγία, για το αν ε, θα έχουμε κάποιες λέξεις ε, όπως το σάλ που ε, μας δείχνουν μέσως ότι έχουμε υποχρεωτικό χαρακτήρα του μέσου και εργαζόμαστε λοιπόν με ένα κείμενο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε έχουμε σύσταση είτε έχουμε οδηγία, δηλαδή είτε έχουμε δεσμευτικό είτε μη δεσμευτικό έγγραφο. Αυτό είναι το εγχείρημά μας. Τώρα, αφήνοντας ε, κατά μέρου τη φύση της νομικής πράξης, σημειώσαμε πρόοδο. Προχωρήσαμε με μια ταχύτητα, αν και προσωρινά έχουν δεθεί τα θέματα, δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουν κλείσει. Ανακαλύψαμε όμως ότι πέρα από δύο-τρία στοιχεία είναι, υπάρχει αρκετά ευρία συνένεση. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το ανέφερα και τώρα με τους εμπειρογνώμονε και εμένα μου προκαλεί μεγάλο λύπη αυτό, ότι υπάρχει μεγάλη, ανθεκτη, μεγάλη αντίρρηση ε, και στη σύσταση 2-3 αλλά και στην αιτιολογική έκθεση όπου αναφέρεται το κύριο στοιχείο από τη δική μου άποψη της πρόβλεψης και της προετοιμασίας για τις τεχνολογικές αλλαγές να δίνεται μία κατάρτιση, δηλαδή μόνιμη για τους εργαζομένους. Πρόκειται για ένα νέο πολιτισμό, πρόκειται για μια οπτική από την Ευρώπη. Δηλαδή να πούμε από τη σκοπιά τη Ευρώπη και στου εργαζόμενου, αλλά και στου επιχειρηματίε ότι πρέπει να προετοιμάζονται γιατί είναι προφανέ ότι λένε ότι σε 20 χρόνια πρακτικά το 90% των εργαλείων που χρησιμοποιούμε σήμερα είτε στι υπηρεσίε, είτε στη βιομηχανία θα είναι πεπαλαιωμένο. Έτσι λοιπόν θα ήταν ευφυέ και από την πλευρά των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων να προετοιμαστούν για ένα μέλο και θα πρέπει να έχουμε διαβίου κατάρτιση και θα πρέπει να προσαρμοστούν και επιχειρήσεις αν θέλουν να συνεχίσουν να επιβιώνουν. Όμω αυτό το θέμα δεν έχει επιληθεί και το να τα θέσουμε στο χαρτί όλα αυτά και να πούμε στα κράτη-μέλη ότι υπάρχει ένα δίκαιο και υποχρέωση ε, για παροχή κατάρτιση από τι επιχειρήσεις και υπάρχει και υποχρέωση από του εργαζόμενου να δέχονται την κατάρτιση αυτή, αυτό θα είναι δύσκολο. Υπάρχουν ε, και δύο θέματα που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Εγώ ελπίζω ότι τη τελευταία λέξη θα είναι θετική, καθώς υπήρξαν ε, και κάποιες ε, αντιρρήσεις ε, στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Στην αρχική μου έκθεση αναφερόταν ένα αριθμητικό στοιχείο, 500 εργαζόμενοι για τις επιχειρήσεις και για τις επιχειρήσεις αναδιάρθρωση 100 εργαζόμενοι. Πολλοί συνάδελφοι θεώρησαν ότι ήταν πολύ μεγάλος αυτός ο αριθμός καθώς ε, δεν κάλυπτε τις πιο μικρές επιχειρήσεις και επίσης ε, κάποιοι θεωρούσαν ότι ήταν πολύ μικρός αυτός ο αριθμός γιατί μέσω ε, των διάφορων ομίλων θα μπορούσαν να παρακάμψουν τις υποχρεώσεις τους οι επιχειρήσεις. Εγώ έλαβα την απόφαση στις συμβαστικές μου να αφήσω αυτό το στοιχείο, να δώσω μια σαφή ένδειξη ότι μιλάμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους μεγάλους ομίλους και τις μεγάλες επιχειρήσεις αναδιάρθρωσης, όμως ε, κάτι που σχολιάσαμε και με τον καθηγητή, εγώ δεν νομοθετώ εδώ, απλώς μιλώ για πολιτικές συστάσεις και αν κάποια στιγμή υπάρξει από την Κομισιόν νομοθετική πρωτοβουλία, υπηρεσίες της Κομισιόν και αυτό είναι σημείο κλειδί επίσης για να είμαστε συνεκτικοί με τις άλλες οδηγίες, για την διαβούλευση των εργαζομένων κτλ. Οι νομικέ υπηρεσίε τη Κομισιόν θα είναι αυτέ λοιπόν που θα προτείνουν την κατάλληλη στιγμή αν έχουμε νομοθέτημα τα κατόφλια και τους αριθμούς. Εγώ ξεκαθαρίζω από την πλευρά μου δεν έχω πρόβλημα να το αφήσω αυτό ανοιχτό, ακόμη και να το ρυθμίσει η εθνική νομοθεσία. Πρέπει να έχουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Α το πει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρωτοβουλία τη. Ε, Όμω, εγώ νομίζω ότι και πάλι μπορεί να υπάρχει διακριτική ευχαίρεια από την πλευρά των κρατών μελών. Αυτό είναι ένα στοιχείο που νομίζω ότι επίση εξαλείφει ένα μεγάλο μέρο των προβλημάτων και προς στιγμή δεν έχουμε προχωρήσει παραπάνω, Πρόεδρε, όμως εγώ νομίζω ότι με αυτό το χρονοδιάγραμμα και με αυτή τη μεθοδολογία, με ένα πολύ επικοδομητικό διάλογο με τους συναδέλφους, νομίζω ότι θα μπορέσουμε αν ε, όλοι είμαστε δεδομένοι να μετακινηθούμε κάπως από την αρχική θέση, αν όλοι θέλουν να κερδίσουν 100% δεν θα υπάρχει συμφωνία, αλλά ναι, θα υπάρξει συμφωνία. Εγώ είμαι ο πρώτος. Δεν μπορώ να πετύχω το 100% αν και κάποια πράγματα θα μου είναι πολύ επώδυνα, γιατί εμένα μου αρέσει να κερδίζω. Euh, Η κυρία Λόπερ Φοντάνια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία με τον κύριο Σέρκας. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να κερδίσουμε. Και γι' αυτό πρέπει να καταλήξουμε στη συμφωνία και να καταλήξουμε στη συμφωνία θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ ακόμη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει με ηρεμία να αναλύσουμε όλο το ζήτημα και κυρίως ό,τι αφορά την πρόβλεψη και τη διαβούλευση αλλά και την ε, κατάρτιση. Αυτά είναι θεμελιώδη σημεία και νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για αυτό το θέμα. Επίσης, θέλω να ζητήσω από τον εισηγητή. Το εξή. Υπάρχει ένα πρακτικό ζήτημα στη σύνταξη των ε, συμβαστικών τροπολογιών. Δηλαδή να διαφοροποιήσετε κάπω ε, περισσότερο του συμβασμού, να υπάρχουν περισσότεροι παράγραφοι, περισσότερες παράγραφες. Δηλαδή γιατί στην ε, συμβαστική πρόταση υπαριθμών 1 έχουμε 33 τροπολογίε. Λοιπόν, είναι πάρα πολλέ οι παράγραφοι και δεν είναι τόσο ευανάγνωστο το κείμενο. Σε ό,τι αφορά τώρα την κατάρτιση και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτής, Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να αναζητήσουμε μια διαφορετική διατύπωση. Γιατί η δική μου ομάδα μπορεί να πιστεύει μένω ότι αυτό είναι ουσιαστικό θέμα, η κατάρτιση. κανεί δεν το αμφισβητεί άλλωστε. Όμω, ο όρος υποχρεωτικό χαρακτήρα είναι κάπω δύσκολο να τη δεκτούμε. Και για τι επιχειρήσει, ε, αλλά και για του εργαζομένου. είναι δύσκολο να δεχτούμε αυτόν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα. Κατάρτιση ναι, αλλά Κοιτάξτε, το υποχρεωτικό χαρακτήρα να το δούμε πώς μπορούμε να το επιλύσουμε. Επίσης, πρέπει να εμβαθύνουμε σε δύο σημεία. Όπως είπαν και οι προσκεκλημένοι και όσοι πήραν το λόγο προηγουμένως, δεν ε, πρέπει να υπάρχουν αντιφάσεις με τη σημερινή νομοθεσία και θα πρέπει να δούμε ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Και τέλος, όπως είπε και ο συνάδελφος Σέρκας, θα πρέπει να αποφασίσουμε με ηρεμία αν θέλουμε στην έκθεση της αναδιάρθρωσης να έχουμε οδηγία ή να μιλάμε για οδηγία για σύσταση. Ξέρετε, η δική μου ομάδα δεν θέλει περισσότερες οδηγίες. Αλλά να το δούμε στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά όμως τη σύνταξη των συμβαστικών προτάσεων, δεν θα έχουμε την ίδια σύνταξη του κειμένου, μιλάμε για δεσμευτική νομοθεσία ή μη δεσμευτική νομοθεσία και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριος Μπενιόν. Μάλιστα. Ε, δεν είμαι ο σκιώτης εισηγητής σε αυτήν εδώ την έκθεση. Την ξεφύλισα αυτό το απόγευμα, να ομολογήσω. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι έφτασα στα βάθη της έκθεσης αυτής, αλλά να αναφέρω δύο πράγματα μόνο. Καταρχάς, πιστεύω ότι έχω κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τη μεθοδολογία και τη χρησιμοποίηση του ίδιου κειμένου, είτε αυτό είναι νομοθετικό είτε όχι. Σίγουρα η ομάδα μας κατέθεσε πολλές ε, τροπολογίες και το ονόμασε ε, κώδικα πρακτικής. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα... Ε, Χαίρομαι πάρα πολύ να δώσω έναν κώδικα δεοντολογίας, αλλά όχι σε μια οδηγία. Ε, πιστεύω πως είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί αυτή η μεθοδολογία, διότι πώς μπορείς να πάρεις μία απόφαση αν θέλεις κάτι, αν δεν θέλεις κάτι, εάν δεν ξέρεις τι αντιμετωπίζεις, σε τι αναφέρεσαι. Και κατανοώ το επιχείρημα του κυρίου Σέρκας ότι εδώ δεν νομοθετεί αυτός, διότι πρέπει να περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Συμβούλιο, να τους ακούσουμε μετά, να επιστρέψει σε εμάς κτλ. Και θα καταλήξουμε κάπου πολύ μακρύτερα από εκεί που έχουμε αρχίσει. Επίσης, συμφωνώ με το σημείο όσον αφορά την κατάρτιση, διότι Καταρχάς, οι εργαζόμενοι διαφόρων τομέων έχουν και διαφορετικές απαιτήσει ε, σχετικά με την κατάρτισή τους. Και δεύτερον, οι απαιτήσει για την κατάρτιση όσον αφορά το πόσες μέρες ε, το χρόνο χρειάζονται ε, διαφέρουν και ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο και από χρόνο σε χρόνο επίσης. Δηλαδή μπορεί φέτος να χρειάζονται πολύ περισσότερη κατάρτιση με καινούργια δεδομένα για έναν εργαζόμενο. Του χρόνου όμως δεν θα χρειαστεί να τον, ε, να του, να τον καταρτήσω για τις ίδιες πολλές μέρες, εάν ισχύουν τα ίδια ίδιες ε, προδιαγραφές. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως εδώ πέρα, εάν μπούμε σε λεπτομέρειες και ονομάσουμε αριθμούς, τότε η βιομηχανία θα έχει αντιρρήσεις και θα μας φέρει ε, μεγάλη αντίρρηση. Θα μας πει πως υπάρχουν και όρια και σταματήστε εδώ. Οι ανάγκες της... Οι ανάγκε των επιχειρήσεων πρέπει να είναι και αυτό κάτι που θα λάβουμε υπόψη μα ε, σε αυτήν εδώ την έκθεση. Επιπλέον, ναι μεν λέμε για επιβράδυνση της διαδικασία αναδιάρθρωσης. Πολύ συχνά όμω, οι αλλαγές στην αγορά γίνονται πολύ γοργά. Και όταν πουλά τα μισά, όταν η εταιρεία σου κάνει τις μισές πωλήσει και έχει 500 απασχολούμενους, μέχρι να τελειώσει η διαδικασία αναδιάρθρωσης θα έχει πέσει έξω και θα έχει χάσει όλε σου τι δουλειέ. Δεν θα έχει μείνει κανένα από του 500. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τι ανάγκε των επιχειρήσεων για ευελιξία και άμεση ανταπόκριση στι αλλαγέ τη αγορά. Διότι μακροπρόθεσμα θα χαθούν πολύ περισσότερε θέσει εργασία εάν είμαστε υπέρ των δέων περιγραφικοί στο πώς ε, και στο πότε και στο πού. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή. Κανονισμός, οδηγία. Δεν έχουμε όμως χρόνο έτσι κι αλλιώς. Αφήστε, αφήστε. Ο εισηγητής ο εισηγητής. Εγώ δεν ζήτησα να πάρει το λόγο η Κομισιόν γιατί είναι πολύ άγουρο ακόμη το ζήτημα, θα πρέπει να οριμάσει. Και κοιτάξτε αυτό το τόσο πράσινο μήλο δεν, ε, δεν είναι και κατάλληλο για την υγεία της Κομισιόν, να σου λίγο. Λοιπόν, τα θέματα που έθεσε η συνάδελφος, η κυρία Λόπε Φορτανιέ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν οι συμβιβαστικέ προτάσει μπορούν να παρουσιαστούν με άλλο τρόπο, θα το πράξω αυτό. Πιθανότατα είναι απλό. Απλώς ε, θα πρέπει να συνδέσουμε τώρα τους συμβασμούς με τις συστάσεις. Για το θέμα της κατάρτισης δεν θα απαντήσω. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο δεν πρέπει να έχουμε επιφυλάξεις. Ε, καταρχήν ε, πρέπει να διαβάσουμε τι λένε εμπειρογνώμες, ποιο είναι το κόστος της κατάρτισης και της μη κατάρτισης. Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι ευφυές, όχι μόνο να θέσουμε και να λέμε πόσο κοστίζει αυτό, αλλά να πούμε και τι θα μας κοστίσει αν δεν το κάνουμε. γιατί την πιθανότητα και λάβαμε και κάποια εξήγηση σήμερα το απόγευμα, είδαμε τι κοστίζει αλλά όχι μόνο σε κοινωνικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο να μην προετοιμάζουμε τους ανθρώπους για τις τεχνολογικές αλλαγές και για την κατάρτιση δεν θέλουμε ουσιαστικά να αναθέσουμε νέο φόρτο στις επιχειρήσεις θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις αν αποτύχουν οι επιχειρήσεις και η κοινωνία αποτυγχάνει και η κοινωνία πρέπει να πει στις επιχειρήσεις ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών, γιατί η εμπειρία μας λέει ότι στο βαθμό λοιπόν που θα το δούμε στο μέλλον. Αλλά αν δεν υπάρχει κάτι που να προέρχεται από τις δημόσιες αρχές, από το κοινοβούλιο, από τα κράτη-μέλη, από τους κοινωνικούς εταίρους που να αλλάξει την κατάσταση, η αδράνεια μας οδηγεί στο 85% των εργαζομένων να μην έχει κατάρτιση. Και αυτό είναι αδύνατο αν θέλουμε η Ευρώπη να συνεχίζει να αποτελεί ένα πρωταγωνιστή σε διεθνές επίπεδο. Εγώ θα συνεχίσω να προσπαθώ να σε πείσω, Βερόνικα, και ουσιαστικά θα πρέπει να αφήσουμε κάθε κράτος μέλος να το ρυθμίσει στο δικό επίπεδο, να το ρυθμίσουν οι κοινωνικοί εταίροι. Αλλά α δείξουμε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη. Την κατεύθυνση, χωρίς ε, να μπούμε σε μια υπερρυθμιστική διαδικασία, δηλαδή να ρυθμίσουμε και τι πιο μικρέ λεπτομέρειε. Σε κάποια τροπολογία αναφέρω και το θέμα τη συνοχή με τι άλλε οδηγίε, αλλά είναι πολύ τεχνικά, πολύπλοκο το ζήτημα. Λοιπόν, ε, εγώ... Κοιτάξτε, δεν μπορείτε να μου ζητάτε σε μια νομοθετική, σε μια τέτοια έκθεση πρωτοβουλία να απαντήσω σε τόσο πολύπλοκα ζητήματα και να προσπαθήσω να λύσω αυτό το πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε εμεί ε, αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι μα ξεπερνάει και θα πρέπει να περιμένουμε να εμφανιστεί κάποια νομοθετική πρωτοβουλία. Για το σου είπε ο κύριο Μπένιον, για τη μεθοδολογία. Κοιτάξτε, να μην μπούμε σε μια ε, συζήτηση νομιλιστική. Κοιτά, εσείς ε, είπατε εδώ ότι θέλετε, ε, αναφερθήκατε σε κάτι δεσμευτικό, όμως ε, δεν υπάρχει σε επίπεδο ο κώδικας ε, των πρακτικών. Υπάρχουν άλλα πράγματα, υπάρχουν πράξεις μη δεσμευτικές, αλλά δεν υπάρχει όρος κώδικας των πρακτικών και πάντα είναι θέμα συνοχής. Στη διάσκεψη των Προεδρών είπαμε ότι ακολουθούμε μια νομοθετική πρωτοβουλία. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στις ε, συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να μην έχουμε ε, δεσμευτικά μέσα. ούτε ή άλλως ούτε οι εμπειρογνώμονες δεν θα μας αφήσουν. Γιατί εδώ μιλάμε για κάτι που δεν υπάρχει. Μίλησα για μήλα εγώ θα ήθελα ένα πάρα πολύ κόκκινο μήλο. Εσείς μπορείτε να μου το ζητάτε πιο πράσινο. Λέω μου ζητάτε χλάδι, γιατί αυτό το δέντρο δεν παράγει. Αχλάδια μήλα παράγει. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι τέτοιο στη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. σε αυτό που σα ανησυχεί είναι το δεσμευτικό ή το μη δεσμευτικό. Θα τη βρούμε τη λύση. Εκτό ε, μικροφώνου το σχόλιο. Όχι, όχι. Εσείς ε, ουσιαστικά υπερβαίνετε και τις ε, μεγαλύτερες επιθυμίες μου. Δεν ανησυχώ. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος, αν δεν πούμε τίποτα, δεν θα κάνουμε βήμα προς τα μπρος. Και τέλος, φροσύνη και ευελιξία. Θα ήθελα εσεί να προβείτε σε μία βάθο ανάγνωση, όχι ταχεία όπω κάναμε τώρα, και να δείτε με πόση προσοχή έχουν γίνει όλα για να μην βλάψουμε τι επιχειρήσει. Όπω ε, υπόθηκε, Θέλουμε ουσιαστικά να πούμε ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί μερικές φορές ε, και η διαδικασία της αναδιάρθρωσης. Ισχύει αυτό, δηλαδή μπορεί να συμβούν πρόβλεπτα κάποια πράγματα γιατί οι αλλαγέ μπορεί να γίνουν ε, λόγω ανωτεράς βίας. Δεν θέλουμε να κάνουμε το δύνατο, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε συνεχώς, να προβλέπουμε τις αλλαγές, ε, αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κερδίσουν το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Κατάλαβα ότι χρειάζεται κι άλλη επεξεργασία των συμβιβαστικών τροπολογιών. Πιστεύω όμως ότι θα βρεθεί η ε, χρυσή τομή. Ευχαριστούμε τον Φιλιππένιο, την κυρία Φοντανιέ και Περιμένουμε τις προτάσεις. Τελειώσαμε με την ημερήσια διάταξη. Στις 6 Νοεμβρίου από τις 3 ως τις 6.30 έκτακτη συνεδρίαση. Μείνετε όλοι μέσα στην αίθουσα. Ελάτε όλοι εδώ. Γιατί σε λίγα λεπτά θα ακολουθήσει συνεδρίαση με τον Επίτροπο στα πλαίσια του διαρθρωτικού διαλόγου. Φέρτε κόσμο όσο πιο πολλούς μπορείτε.